Control me, please. Yes. So, ladies... Κυρίες και κύριοι. Κυρίες και κύριοι. Καλωσορίζω όλους σας. Και επιτρέψτε μου να ξεκινήσουμε τις σημερινές μας εργασίες. Μαρκρέτε. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε τις σημερινές μας εργασίες. Να ρωτήσω, υπάρχουν ε, αντιρρήσεις ως προς την ημερήσια διάταξη. Όχι. Εγκρίνεται λοιπόν η ημερήσια διάταξη. Έχουμε δύο σειρές πρακτικών ε, από τον Νοέμβριο και τον Ιανουαρίου. Δεν έχουμε λάβει καμία αντίδραση. Όντως, ωραία, εγκρίνονται λοιπόν τα πρακτικά. Δεν υπάρχουν ε, ανακοινώσεις του Προέδρου και τα διάφορα θα συζητηθούν στο τέλος της ενής συνεδρίασης, μάλλον ο Πέδρος. Ε, να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Έχετε τις κάρτες σας. Άρχεται η ψηφοφορία. 4, 3, 2, 1... Ξεκινάμε λοιπόν. Συμβαστική 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 30. Υπέρ. In, in favor. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. So now 32. 32. Amendment 32 in favor. Τροπολογία 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 της ηγήτριας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση. The vote is closed. Άρχεται η ψηφοφορία, λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται σαφώς. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 5 και 11 υπέρ κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνονται. Τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία ονομαστική. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 14 ψήφου υπέρ. Σας ευχαριστώ πολύ. Λίγη ψηφοφορία. Okay. Please, I would like to continue in our program. Να συνεχίσουμε λοιπόν τώρα στην ημερήσια διάταξή μας. Ένα λεπτό. Διακοπή για τεχνικούς λόγους. So I would like to change the language Θα ήθελα να μιλήσω σλοβακικά. Κυρίες και κύριοι, περνάμε στη συζήτηση για την διαρευνητική επίσκεψή μας στο Εθνικό Πάρκο Τονιάνα της Ανταλουσίας. Ήμουν εγώ πρόεδρος ε, της αποστολής και θα ήθελα να σας ενημερώσω σχετικά με την επίσκεψή μας εκεί. Το Εθνικό Πάρκο της Ντονιάνα είναι πολύτιμο για την Ευρώπη. Είδαμε κατά τη διάρκεια της επίσκεψή μας σε πολλά θετικά μέτρα που έχει αναλάβει η Ισπανία. Υπάρχουν κάποια προβλήματα και μάλιστα διτής φύσης στο πάρκο αυτό τις τελευταίες δεκαετίες σε κάποιες ζώνες είχαμε παραγωγή αερίου. Η αποθήκευση του αερίου δημιούργησε κάποια προβλήματα. Το συζητήσαμε αυτό με τους επικεφαλείς του πάρκου με τη διεύθυνση του πάρκου και με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. συμπεριλαμβανομένης ε, της εταιρεία που είναι αρμόδια για την υποδομή. Συζητήθηκε και η πιθανότητα σεισμών στο πλαίσιο αυτό. Την έκθεση της επίσκεψής μας ε, μπορείτε να τη βρείτε στα έγγραφά σας. Μπορούμε λοιπόν ε, στις προθεσμίες μέχρι τις 4 Μαρτίου μπορείτε να υποβάλλετε σχετικές προτάσεις για την έκθεση αυτή. 4 Μαρτίου στις 3 λοιπόν είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Η έκθεση αυτή έχει συνταχθεί μετά από την επίσκεψή μας στην Ισπανία. Προχωράμε στην συζήτηση πάνω στο θέμα αυτό και θα ήθελα καταρχάς να δώσω το λόγο στον Δανιέλ Φερνάντες Κόμες, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κρατά την Επιτροπή σας ενήμερη σχετικά με οποιασδήποτε νέες πληροφορίες λάβουμε σχετικά με την αναφορά για το πάρκο Ντονιάνα καθώς και για τις αναφορές που έχουν να κάνουν με την παραγωγή και αποθήκευση φυσικού αερίου καθώς ε, και τις αιτήσει ε, που έχουν να κάνουν με τον ε, με τον υδροφόρο ορίζοντα. Υπήρχε αναφορά για την παραβίαση της οδηγίας για τα ύδατα, της οδηγίας πλαίσιο, καθώς και για την καταστροφή των φυσικών οικοτόπων. Ζώνες Natura 2000 στο Πάρκο Ντονιάνα, καθώς και σε γειτονικές περιοχές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή συγκεντρώνει τα έγγραφα για την υπόθεση και θα εναπόκειται στο δικαστήριο να αποφασίσει εάν η, Ισπανία ε, τηρεί τις υποχρεώσεις της ε, σύμφωνα με τις οδηγίες που ανέφερα. Όσον αφορά τα υπόλοιπα έργα, όπως ε, ήδη έχω πει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει διαπιστώσει καμία παραβίαση του ενωσιακού δικαίου. Έχουμε ζητήσει από τις Ισπανικές Αρχές ε, να μας κρατούν ενήμερους ε, σχετικά με οποιοδήποτε νέο γεγονός μπορεί να επηρεάσει τα προγράμματα αυτά. Η Επιτροπή θα κρατήσει ενήμερη την Επιτροπή σας σε περίπτωση που λάβουμε νέες πληροφορίες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Η κυρία Αλμπίολ έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την όλη εργασία που κάνατε, για τη σύνταξη της έκθεσης αυτής. Θα είχαμε θελήσει να τη λάβουμε λίγο νωρίτερα, γιατί έχουν μεσολαβήσει πέντε μήνες από τότε που πήγατε στην Τονιάνα που πήγαμε μάλλον στην Τονιάνα και νομίζω ότι θα έπρεπε και τα υπόλοιπα μέλη να μπορούν να ενημερωθούν εγκαίρως πιο γρήγορα για το ζήτημα αυτό. Τώρα όσον αφορά το περιεχόμενο αυτό καθεαυτό εν γέννη, θεωρούμε ότι ε, η έκθεση δεν είναι ιδιαίτερα φιλόδοξη. Δίδεται η εντύπωση ότι η έκθεση αυτή συντάχθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να μην ενοχλήσουμε πολύ τις ισπανικές αρχές. Παρ' όλα αυτά, οι Ισπανικές αρχές είναι οι πλέον υπεύθυνες για την τρέχουσα κατάσταση στο Εθνικό Πάρκο Ντονιάνα. Και δυστυχώς δεν γίνεται σχετική αναφορά στην έκθεση αυτή. Δεν λέγεται ξεκάθαρα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει συγκεκριμένα μέτρα κατά της Ισπανίας. Μόλις τώρα το είπε ο πρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο οποίο είπε ότι θα μπορούσε να οδηγηθεί ακόμα και στο δικαστήριο η Ισπανία, επειδή οι ισπανικέ αρχές δεν λάβαν τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσουν το Εθνικό Πάρκο της Ντονιάννα. Θα θέλαμε λοιπόν η έκθεση να λέει αυτό το στοιχείο. Επίσης, πρέπει να στηρίξουμε το τι έχουν κάνει μέχρι στιγμής οι αρμόδιες αρχές. Γιατί αυτά που έχουν γίνει μέχρι στιγμής είναι αυτό το οποίο οδήγησε στη σημερινή κατάσταση στη Τονιάνα. Είναι δηλαδή στο να είναι στον κατάλογο των επικίνδυνων περιοχών της UNESCO. Και αυτό που μας σχολίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, ε, το σχέδιο της έκθεσης είναι πάρα πολύ ε, ανισόρροπο ως προς τις απειλές. Ε, ως προς την προστασία των, α, α, των υδάτινων πόρων ε, δεν είναι μόνο η εκμετάλλευση του υδροφόρου ορίζοντα το πρόβλημα. Μόνο μία από τις δύο συστάσεις μιλάει για την απειλή ότι μπορεί να γίνει η Ντονιάνα μία αποθήκη φυσικού αερίου. Υπάρχουν πάρα πολλές ε, αναφορές οι οποίες μιλούσαν για το πρόβλημα της αποθήκευσης ε, φυσικού αερίου ε, στην Τονιάνα. Δεν είναι λοιπόν μόνο το πρόβλημα των υδάτινων πόρων. Θα πρέπει να βάλουμε και το θέμα της αποθήκευσης φυσικού αερίου. Επίσης, το γεγονός ότι η έκθεση μιλάει για την σημασία της αρχής της πρόληψης και της προφύλαξης και θα πρέπει να γίνει μια περιβαλλοντική μελέτη για να δούμε τους κινδύνους για σεισμούς είναι πάρα πολύ θετικό. Και είναι θετικό το ότι αναφέρει η έκθεση. Αλλά νομίζουμε, νομίζουμε ε, ότι η μόνη πραγματική πρόληψη είναι να σταματήσει ε, οριστικά αυτή η διαδικασία εξόριξης φυσικού αερίου στην Τονιάνα. Ε, Υπάρχουν οι τροπολογίε λοιπόν που θα υποβάλουμε για την έκθεση, ούτω ώστε να φτιάξουμε τελικά μία έκθεση που θα μας ε, οδηγήσει στις κατάλληλες συστάσει για να προστατεύσουμε την Τονιάνα. Ευχαριστούμε πολύ. Να πω απλώς συναδέλφους ε, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κινήσει τη διαδικασία παραβάση κατά της Ισπανίας στα τέλη Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους και νομίζω ότι θα μας είχε βοηθήσει όλος ιδιαίτερος κατά τη διάρκεια της διερευνητικής επίσκεψης να είχαμε τις πληροφορίες αυτές γέρος. Καταρχάς να σας πω ότι η Ντονιάνα έχει τεράστια αξία. Είναι στοιχείο της ταυτότητάς μας και για την Ουέλβα, για την Ανδαλουσία και για όλη την Ισπανία τελικά. Και η διατήρησή της είναι ένας στόχος δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι έτσι τα πράγματα και ειδικά είναι πολύ πιο σημαντικό για τους ανθρώπους που ζουν στην περιοχή ή πιο κοντά στην περιοχή. Με, αυτή την, με αυτά που μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμείς θέλουμε να τονίσουμε το πρόβλημα των υδάτινων πόρων για να διατηρήσουμε και να σεβαστούμε αυτή την κληρονομιά δεν αμφιβάλλω ότι πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα από τις αρχές. Αυτό νομίζω ότι έλαβε υπόψη της Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν έκανε αυτή την προσφυγή. Ε, υπάρχει αυτό το σχέδιο του, της Κορούνια του Βορρά και η τοπική κυβέρνηση της Ανδαλουσίας επί χρόνια δεν έκανε τίποτα. Ε, πριν από ένα μήνα άρχισε να κάνει κάποια πράγματα υπέρ του νερού και γίνανε κάποιες επικαιροποίησεις ε, του σχεδίου αυτής, αυτού. Υπήρχε λοιπόν αυτή η ανησυχία και υπήρχε μια απόπειρα να δοθούν απαντήσεις στις απειλές. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι υπάρχει υπερεκμετάλλευση γεωργικής φύσεως. Είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε ότι αυτή η υποτιθέμενη ε, υπερεκμετάλλευση που σε γεωργικό επίπεδο είναι πολύ σημαντική και για λόγους κλιματικής αλλαγής. Όταν γίνεται υπερεκμετάλλευση γεωργική, έχουμε υπερβολική χρήση του νερού, αλλά πρέπει να το βάλουμε αυτό μέσα σε ένα πλαίσιο. Ε, αυτό το πάρκο είναι εθνικό πάρκο, είναι μια μικρή ζώνη, πρέπει να έχουμε ένα πλαίσιο σωστό. Και μετά υπάρχει ε, μια άλλη μεγαλύτερη ζώνη με διαφορετική διαβάθμιση προστασίας. Αυτό το φυσικό ε, πάρκο όλο και μεγάλωνε, ναι, ενώ υπάρχουν συγκεκριμένες οικονομικές πραγματικότητες στην περιοχή. Μην ξεχνάμε ότι χρειάζεται η γεωργία ε, στην περιοχή. Δεν αρνούμε ότι υπήρξε υπερεκμετάλλευση, αλλά υπάρχει μεγάλο θέμα οικονομικό στην περιοχή. Πρέπει να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή. Όταν λοιπόν ε, εκτοξεύουμε κατηγορίε, να λάβουμε υπόψη μα και την οικονομική διάσταση. Ναι, να διατηρήσουμε την προστασία τη Ντονιάνα, αλλά να μην ξεχνάμε και τι υπόλοιπε πραγματικότητε, οικονομικά κτλ. Το 2016 είναι η τελευταία έκθεση που έχουμε ε, για την Ντονιάνα από την UNESCO. Από ε, την UNESCO. Αναφερόταν αυτέ οι απειλέ, αλλά αναφερόταν ότι είχαν ξεκινήσει οι αρχέ τα αρμόδια μέτρα για να επιληθούν τα προβλήματα. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διατηρήσουμε την περιοχή. Πιστεύω ότι το θέμα του φυσικού αερίου είναι σημαντικό, πρέπει να το τονίσουμε περισσότερο, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Αλλά άκουσα αυτό που μου είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν υπάρχει παραβίαση, έτσι. Σημαντικό αυτό. Μην ξεχνάμε ότι έγινε μελέτη περιβαλλοντικής επίπτωσης και εκεί διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει παράβαση. Τέλος. Πέρα από τις απειλές. Νομίζω ότι πρέπει να φτιάξουμε μία έκθεση που να έχει θετικό τόνο. Γιατί νομίζω ότι συνηθίζουμε να μιλάμε έτσι πολύ άσχημα. Ε, εντάξει, μιλάμε για μία περιοχή, για μία επαρχία, ας πούμε, που έχει μία ζώνη προστατευόμενη. Αλλά μην ξεχνάμε από την άλλη και την οικονομική διάσταση, την οικονομική ανάπτυξη. Ε, μην ξεχνάμε, δηλαδή, τι συμβαίνει γύρω-γύρω από την Τονιάνα. Πρέπει να κάνουμε θετικές προτάσεις στην έκθεσή μας. Γιατί αν θέλουμε να διατηρήσουμε το περιβάλλον και να το αξιοποιήσουμε, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και την οικονομική διάσταση, την οικονομική αξία που έχει το περιβάλλον, έτσι. Που μην ξεχνάτε ότι η ακτή της Σουέλβα είναι η μόνη ακτή της Ανταλουσίας που είναι ανεπτυγμένη. Συγγνώμη, που δεν είναι ανεπτυγμένη και θα πρέπει να την αναπτύξουμε. Πέρυσι έγινε πυρκαγιά στην Τονιάνα, σε αυτό το πάρκο που θέλουμε να υπερασπιστούμε δεν υπήρξε καμία βοήθεια οικονομική για την αναδάσωση της περιοχής αυτής από την Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή. Είναι μια περιοχή ειδική, προστατευόμενη. Πρέπει να αξιοποιήσουμε το περιβάλλον και οικονομικά να το αξιοποιήσουμε ενώ, ούτω ώστε να το προστατεύσουμε τελικά. Αν αξιοποιηθεί, προστατεύεται. Γιατί αυτή η φυσική περιοχή, η προστατευόμενη περιοχή, έχει και μία οικονομική αξία και αυτή πρέπει να τη λάβουμε υπόψη μας. Eh, αυτή η έκθεση πηγαίνει προς σωστή κατεύθυνση, νομίζω. Χάρη και στις κοινωνικές πιέσεις των κατοίκων της Ντονιάνα και της Ανδαλουσίας, έγινε μια καλή δουλειά τελικά, ούτω ώστε να μπει το θέμα της Ντονιάνα σε μια πορεία μεγαλύτερης βιωσιμότητας περιβαλλοντικής και κοινωνικής. Αυτή η έκθεση βεβαίως έχει κάποιες ελλείψεις και είναι κάπως άτολμη, θα μπορούσε να είναι πιο σαφής ας πούμε. Ορισμένα πράγματα λέμε αμφισημεία. αμφισημία, θα, θα μπορούσε να τα πει πολύ πιο σαφώς. Μερικές φορές, ας πούμε, τονίζουμε υπερβολικά το θέμα της ε, ξηρασίας. Όχι, εγώ νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα νερού, γιατί ε, παίρνουμε νερό, σκάβουμε πηγάδια, ας πούμε, παίρνουμε νερό για να το χρησιμοποιήσουμε για τη γεωργία. Υπάρχει αυτό το ειδικό σχέδιο για την Τονιάνα από το 2014 καταγράφει 2.500 πηγάδια ε, εξόριξης για νερού. Πολλά από αυτά μάλιστα είναι παράνομα. Είναι χίλια τα μη ε, επιτρεπόμενα πηγάδια. Τα παράνομα πηγάδια που έχουν ε, δημιουργηθεί. Και η ίδια η τοπική κυβέρνηση αναγνωρίζει αυτή την πραγματικότητα. Πέρα από αυτά που μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει ανοίξει διαδικασία εναντίον της, ε, των αρχών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. θα πρέπει να είναι πολύ πιο σοβαρή η διαδικασία που κοινή Επιτροπή, γιατί υπάρχουν ε, αυτά τα παράνομα πηγάδια που δεν λαμβάνονται υπόψη στην ε, διαδικασία. Υπάρχει λοιπόν το θέμα του νερού, που το συζητήσαμε, και υπάρχει και το θέμα του φυσικού αερίου. Ακριβώς για το φυσικό αέριο πήγαμε στην Τονιάννη και κάναμε την επίσκεψη. Επίσης, δεν μπορούμε να κάνουμε σχέδια ε, μεμονωμένα. Θα πρέπει να έχουμε ένα συνολικό σχέδιο. Επίσης θα θέλαμε η Ισπανική κυβέρνηση να μας πει με ξεκάθαρο τρόπο ότι αυτή, αυτό το σχέδιο για την εξόρυξη φυσικού αερίου δεν είναι στρατηγικού χαρακτήρα. Πρέπει να το πει. Δεν, έχει, δεν γίνεται για το, καλό, για το κοινό καλό αυτό το project. Θα πρέπει να τονιστεί αυτό το στοιχείο και στην έκθεση. Θα ήθελα τώρα να τελειώσω με ένα διαδικαστικό θέμα γιατί με ενοχλεί πάρα πολύ. Η κλασική πρακτική είναι να ξεκινήσουμε την ε, ε, έκθεση και να δώσουμε χρόνο στα μέλη, ούτως ώστε να υποβάλουν ε, παρατηρήσεις. Εγώ δεν είχα χρόνο να υποβάλω τις παρατηρήσεις μου. Δεν είχαμε χρόνο. Δεν μπορούμε λοιπόν να το επιτρέψουμε αυτό. Δεν είναι σωστό αυτό. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γίνεται αυτό. Θέλω εξηγήσει λοιπόν. Γιατί ζητώ λίγο σεβασμό. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Φεραγκούτ για την προθεσμία για τις τροπολογίες. Ε, είναι σημαντικό αυτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σάκη και τα άλλα μέλη που ετοίμασαν αυτή την έκθεση. Νομίζω ότι θα πρέπει να κρατήσουμε αυτές τις πληροφορίες που μας έδωσε η Κομισιόν και να ξεκινήσουμε ε, για το θέμα των, του υδροφόρου ορίζοντα ε, διαδικασία ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Για τα παράνομα πηγάδια θα πρέπει να το δούμε ε, αυτό το θέμα. Κάναμε μια συνεδρίαση όπου ήρθαν οι Γεωργοί και μιλούσαν ε, για, τα παράνομα πηγάδια. Αλλά μας είπαν ότι δεν είναι σωστό να τιμωρήσουμε γι' αυτό ε, όλους τους ε, γεωργούς, γιατί δεν έχουν όλοι παράνομα πηγάδια. Νομίζω και εγώ λοιπόν ότι πηγαίνουμε προς την σωστή κατεύθυνση και το άλλο θέμα για το θέμα του φυσικού αερίου. Το μόνο πρόβλημα που βλέπω και μας το είπε και ο εκπρόσωπος της τοπικής κυβέρνησης είναι ότι πολλές, τοπι... πολλές ε, ανδαλουσιάνικες αρχές και ισπανικές αρχές ε, δεν έχουν ε, τη συνολική εικόνα για όλες τις άδειες κτλ. Πρέπει να υπάρχει ασφάλεια δικαίου. Ούτως ώστε να μην υπάρξουν ε, πολλές αμφισβητήσεις για άδειες που έχουν δώσει διαφορετικές αρχές. Πρέπει να κάνουμε διάφορα πράγματα. Να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια δικαίου, ε, να προστατεύσουμε το περιβάλλον και τη σημασία που έχει η τοποθεσία αυτή, αλλά να τη συνδυάσουμε με τις γεωργικές δραστηριότητες που υπάρχει από πάντα. Γιατί ε, και χάρη στους γεωργούς διατηρήθηκε το πάρκο στην κατάσταση. Δηλαδή, διατηρήθηκε. Είναι σημαντική η, συμβολή τους. Πιστεύω ότι με τις α, τροπολογίες θα βελτιώσουμε περισσότερο τα, τις απόψεις του κυρίου Σάκη, αλλά ήδη τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Μιράντα, στη συνέντευξη τύπου η Κομισιόν μας είπε ότι έχει ανοίξει διαδικασία επί παραβάση. Υπάρχει και μια άλλη περίπτωση για το ατύχημα στο Τριγκάνκε, που επίσης ξεκινάει η διαδικασία επί παραβάση. Το είπε η Επίτροπος. Όχι, δεν το κάνουν για πλάκα η Κομισιόν. Ε, επί πολλά χρόνια δεν έγινε τίποτα από τις αρχές. Και τώρα η Κομισιόν προχωράει σε αυτή τη διαδικασία. Δεν καταλαβαίνω ποια είναι η έκπληξή σας λοιπόν, γιατί βλέπω ας πούμε την τοποθέτηση του κ. Μαρθελέση. Ε, δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιοι συναδελφοί είχαν την έκθεση στα χέρια τους και κάποιοι άλλοι. Είναι, δεν είναι σωστό. Δεν είναι η διαδικασία αυτή. Κάποιο μέλος, ας πούμε, ε, της Επιτροπής μας ε, παίρνει στα χέρια του την έκθεση πολύ νωρίτερα από τους υπόλοιπους. Δεν είναι σωστό. Να μας πει η γραμματεία γιατί συνέβη αυτό. Ή θα μας αντιμετωπίζετε όλους με τον ίδιο τρόπο και θα έχουμε πρόσβαση για όλα τα έγγραφα ε, την ίδια στιγμή, ή αλλιώς θα υπάρχουν τα μαύρα πρόβατα. Αλλιώ, αν θέλετε να μπούμε σε άλλα ας πούμε, νομικά επιχειρήματα, ας πούμε, και να πάμε το θέμα στο Προεδρείο. Ή θα μας ενημερώνετε την ίδια χρονική στιγμή όλου, Γενικά τα πράγματα λειτουργούν καλά. Μέχρι τώρα δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Δεν καταλαβαίνω γιατί το είπε αυτό ο συνάδελφο, Με εντυπωσιάζει αυτή η διατύπωση, η διακήρυξη αυτή. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο. Θέλουμε να μάθουμε τι συνέβη ακριβώς. Αγγελάρα, Ευχαριστώ Αγγιλάρ. Υπόθηκαν πάρα πολλά πράγματα. Να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα. Υπάρχουν κάποιες ανακρίβειες για την Τονιάννα και τη λειτουργία της. Ορισμένοι είπαν ότι υπάρχουν διαφορετικές φάσεις του project. Η εθνική κυβέρνηση με πρόεδρο το Ραχώη του ΕΛΚ είναι υπεύθυνο για τις διαφορετικές φάσεις του σχεδίου. Κανένας από τους Ανδαλουσιάνους δεν, δεν θέλησε ποτέ από τι αρχέ Ανδαλουσίας δεν έκανε τίποτα. Ε, ε, ή μάλλον, δεν είναι συνυπεύθυνη η κυβέρνηση Ανδαλουσίας, κυβερνηση ανδαλουσία, μπορεί να θεωρηθεί συνυπεύθυνη με την εθνική κυβέρνηση του ΕΛΚ. Αλλά όχι, δεν έχει καμία ανάμειξη. Ευχαριστώ πολύ. Δεν φαίνεται να ζητάει κανείς άλλο το λόγο. Θα ήθελα λοιπόν να κλείσουμε το θέμα αυτό. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους. και τους συναδέλφους που συμμετείχαν στην αποστολή στην Ισπανία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τη Γραμματεία, διότι ήταν πολύ καλά προετοιμασμένη η επίσκεψη. Δεν ξέρω ποια κείμενα έχουν κυκλοφορήσει. Πάντως μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν ε, υποβλήθηκαν προτάσεις οι οποίες να μην συμπεριληφθούν στο κείμενο. Ε, εγώ ο ίδιος έχω εκπονήσει την έκθεση, μίλησα και με τον κύριο Κύρκο και συμφωνήσαμε όσον αφορά το, τελευταίο, το τελικό κείμενο και αυτό ισχύει. Επαναλαμβάνω λοιπόν. Μπορείτε να υποβάλλετε τις προτάσεις σας, δυστυχώς μόνο στα αγγλικά, μέχρι τις 4 Μαρτίου, στις 3 η ώρα το απόγευμα. Μπορείτε δηλαδή ακόμη να συνεισφέρετε στην έκθεση αυτή να συμβάλλεται στην τελική της διαμόρφωση μέχρι στις 4 Μαρτίου στις 3 ώρα το απόγευμα. Συνολικά είναι η τρίτη αποστολή στην Ισπανία ε, υπό τη δική μου ηγεσία και ε, έχω μια πολύ καλή αίσθηση. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ε, λάβει υπόψη τις σοβαρά τις προτάσεις μας και υπάρχει διάλογος με τις Ισπανικές αρχές. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να βοηθήσουμε την κατάσταση και να τη βελτιώσουμε παρότι γνωρίζω ότι η Βυρική Χερσόνησος έχει επηρεαστεί πολύ από την αλλαγή του κλίματος και έχει όλο και λιγότερο νερό. Αυτό βέβαια δεν είναι πρόβλημα το οποίο να μπορούμε να λύσουμε εμείς εδώ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πάντως όλους και σας καλώ μέχρι τις 4 Μαρτίου, 3 η ώρα, να υποβάλλετε τις τροπολογίες σας. Διακόπτουμε λοιπόν εδώ τον διάλογο στο θέμα αυτό, αλλά θα επανέλθουμε. Σας ευχαριστώ πολύ και περνάμε τώρα στην ε, αναφορά 1088. Δεν έχω το όνομα του αναφέροντος, JR ε, γράφει μόνο, γαλλικής ηθαγένειας. Και το θέμα αυτό αφορά τη, τον νόμο των ε, ΙΠΑ περί φορολογικής συμμόρφωσης αλλοδαπών λογαριασμών, ΦΑΤΚΑ. Με ενημερώνω ότι είναι παρόν ο αναφέρον. Είναι? Ναι, ωραία, καλώς ήρθατε. Σας δίνω το λόγο για πέντε λεπτά. Thank much, Mr. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα χρησιμοποιήσω τα 5 αυτά λεπτά συνοψίζοντας λίγο τα όσα έχουν συμβεί από τότε που παρουσίασα πριν από δύο χρόνια, τον Ιούλιο του 2017, για πρώτη φορά την αναφορά μου σε ένα ζήτημα το οποίο είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο, σαπουνόπερα θα μπορούσαμε να το αποκαλέσουμε κιόλα. Τι συνέβη λοιπόν από τον Ιούλιο του 2017 μέχρι σήμερα. Ο καθηγητής κύριος Γκαρμπαρίνο εξέδωσε μία έκθεση όσον αφορά του νέου κανόνε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίω τον κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τον γενικό κανονισμό GDPR δηλαδή, και αν αυτό μπορεί να συνδυαστεί με τον νόμο των ΗΠΑ περί φορολογική συμμόρφωση αλλοδαπών λογαριασμών. Συζητήσαμε επίση με εμπειρογνώμονε από το Νομένο Βασίλειο που είπαν ξεκάθαρο ότι δεν συνάδουν τα δύο κείμενα. Η πράξη των ΗΠΑ με το GDPR είναι δύο ασύμβατα κείμενα. Ακόμα και αν επιμείνει τελικά η Αμερική στο σύστημα φορολογίας με βάση τους πολίτες και αν συνεχίσει να φορολογεί τους μη μόνιμους κατοίκους τελικά, τότε δεν θα λάβει πραγματικά χρήματα στον δημόσιο κορβανά. Δεν πρόκειται να καταφέρει να φορολογήσει τελικά πολίτες. Τι θέλει να πετύχει λοιπόν μέσω του ΦΑΤΚΑ η Αμερική. Θέλει ουσιαστικά να γνωρίζει περισσότερα πράγματα για τους Αμερικανούς πολίτες που ενδεχομένω να κρύβουν χρήματα στο εξωτερικό. Γι' αυτό ακριβώ το λόγο θεσπίστηκε τελικά αυτή η πράξη φορολογική συμμόρφωση των ξένων λογαριασμών. Μα το τονίζει αυτό ο καθηγητή Καρμπαρίνο και πάρα πολλοί το παραμελούν αυτό, ότι αυτό είναι το βαθύτερο αίτιο, αν θέλετε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους ευρωβουλευτές, οικία πλέον πρόσωπα, να τους ευχαριστήσω για την ε, υποστήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια. Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι ε, στις 5 Ιουλίου του 2018 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα ψήφισμα υπέρ των Αμερικανών λόγω συγκυριών, ένα ψήφισμα που υπερψηφίστηκε με 470 ψήφους υπέρ. Δεν θέλω να επαναλάβω τώρα όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία ήδη τα γνωρίζετε, καθότι και εσείς συζητήσετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το ζήτημα αυτό. Κάναμε σίγουρα πολλέ συζητήσει με εκπροσώπου Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βλέπω ότι υπάρχουν και εκπρόσωποι εδώ πέρα που έχουν έρθει και του γνωρίζω. Και θα έλεγα ότι πολύ συχνά πολύ κρύβονται πίσω από δικαιολογίε. Μην το πάρετε αυτό προσωπικό, αλλά πολύ συχνά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μα λέει δεν γνωρίζουμε τι κάνουν οι πολιτείε με τη ΦΑΤΚΑ, δεν γνωρίζουμε τι κάνουν οι κυβερνήσει κ.ο.κ. Εγώ μεγάλο πολίτη και έχω προσπαθήσει να αναζητήσω πληροφορίε. Έχω και την Ιρλανδική υπηκότητα, απευθύνθηκα και στην Ιρλανδία. Η γυναίκα μου είναι από τη Βρετανία, ζητήσαμε και από εκεί πέρα πληροφορίε. Και σε όλε αυτέ τι αιτήσει πληροφοριών που κάναμε και ενημέρωση, είχαμε αρνητική απάντηση από όλε αυτέ τι κυβερνήσει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι από τη μια μα λένε ότι το ΦΑΤΚΑ υπάρχει για να αυξήσει τη διαφάνεια και από την άλλη δεν υπάρχει καμία διαφάνεια όταν εμεί ζητάμε περαιτέρω ενημέρωση. Και το θέμα είναι ότι οι ευρωπαϊκέ κυβερνήσει γνωρίζουν ότι δεν παίρνουν καθόλου στοιχεία από τι ΗΠΑ, ενώ οι ίδιε δέχονται να διαβιβάσουν τεράστιε πληροφορίε προ τι ΗΠΑ. Μάλιστα, ήρθα και σε επαφή με αρχέ του Καναδά και της Αυστραλίας και προσπάθησαν να δω τι γίνεται με τις χώρες αυτές. Από το 2016 και μετά, από τότε που άρχισε να ισχύει αυτός ο νόμος, ουσιαστικά έχουμε περίπου 18 εκατομμύρια λογαριασμούς, οι πληροφορίες των οποίων έχουν πάει προς τις ε, Ηνωμένε Πολιτείε. Και θα έλεγα ότι 2.400 δισεκατομμύρια ευρώ, αυτό είναι το ποσό στο οποίο αντιστοιχούν όλα αυτά τα τραπεζικά δεδομένα τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προωθήσει προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν αυτό δεν αρκεί για να σας πεις, πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να σας πω. Επίση, εγώ από το 2012 και μετά έχω έρθει σε επαφή με πάρα πολλού ανθρώπου σα έχω κουράσει ενδεχομένω, έχω γίνει φορτικό με όλα αυτά τα email τα οποία στέλνω. Ξέρω ότι υπάρχει επίση το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όσον αφορά την προστασία των δεδομένων και από ό,τι μου είπανε και αυτό μου προκάλεσε εντύπωση, δεν γνωρίζουν οι ίδιοι αυτός ο αρμόδιος οργανισμό, του Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασία Δεδομένων αν τελικά το GDPR και το FATCA μπορούν να συνδυαστούν ως κείμενα. Αν ε, ο νόμος αυτός των ΗΠΑ συμμορφώνεται τελικά με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας των ε, Προσωπικών Δεδομένων. Αυτό πραγματικά με εξέπληξε και ερχόμενο σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησα περισσότερα δεδομένα, λέγοντας ότι ενδεχομένω να υπάρχει παραβίαση των προσωπικών δεδομένων κάθε φορά που διαβιβάζονται τραπεζικά στοιχεία των Ευρωπαίων πολιτών προς ΗΠΑ. Το πρόβλημα είναι ότι ε, οι πληροφορίες αυτές δεν φτάνουν τελικά σε εμά, δεν γνωρίζουμε ποιες πληροφορίες μας διαβάζονται προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και ουσιαστικά θεωρώ ότι εδώ πέρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα υπόλοιπα αρμόδια όργανα τελικά εθελοτυφλούν. Ας μην ξεχνάμε ότι το πρώτο πρόστιμο το οποίο υποβλήθηκε στα πλαίσια του GDPR είναι από την Γαλλική Εθνική Επιτροπή Πληροφορίας Ατομικών Ελευθεριών, το γαλλικό ΚΝΙΛ, το οποίο επέβαλε πρόστιμο 50 εκατομμυρίων ευρώ στην Google. Αυτό που θα ήθελα να σας πω είναι ότι οι τράπεζες θα περιέλθουν σε μια ιδιαίτερα δυσχερή σχέση με τον ΦΑΤΚΑ και νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι το μορατόριουμ, το τελεσίγραφο ουσιαστικά το οποίο έχει τεθεί από τις Αμερικανικές αρχές προς τις Ευρωπαϊκές αρχές για να υποβληθούν στοιχεία που έχουν να κάνουν με τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης κτλ. τελειώνουν στα τέλη του έτους. Τι θα γίνει με ανθρώπους σαν και εμένα ουσιαστικά θα έχουμε εδώ πέρα μια κατάσταση ανάλογη με την επιλογή της Σόφη. Καταλαβαίνετε ότι είτε θα πρέπει ουσιαστικά να προχωρήσουν οι αρμόδιες αρχές σε μια τεράστια παραβίαση των προσωπικών δεδομένων των Ευρωπαίων πολιτών στέλνοντας πάρα πολλά στοιχεία στις ΗΠΑ ή θα πρέπει να αποφασίσουν οι αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές και οι τραπεζικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παραβιάσουν τελικά τον ίδιο τον ΦΑΤΚΑ και να μην στείλουν τα δεδομένα αυτά προς τις ΗΠΑ. Νομίζω λοιπόν ότι αντιμέτωποι με τα νέα αυτά δεδομένα, ίσως την τελευταία στιγμή να αποφασίσετε να μας προστατεύσετε. Αυτό ακριβώς αισθάνονται οι Ευρωπαίοι πολίτες που έχουν και την Αμερικανική ηθαγένεια. Τώρα, πώς εξελίσσονται κατά την άποψή μα τα πράγματα. Θεωρώ ότι μας εξεπλήσει το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασκεί πίεση στις ΗΠΑ όταν τη συμφέρει. Το έχει κάνει αυτό με το υπολογιστικό νέφος, το έχει κάνει με πολλές άλλες πρόσφατες πρωτοβουλίε των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόσφατα πήλησε τις Ηνωμένε Πολιτείε να τις εντάξει στον μαύρο κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους φορολογικούς παραδείσου. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να εμπνευστεί λίγο περισσότερο από τον Καναδά που έχει δείξει πολύ πιο ισχυρή στάση και πυγμή απέναντι στι ΗΠΑ. Η Γαλλία αρχίζει σιγά σιγά να ορθώνει το ανάστημά τη. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει και κάτι από ευρωπαϊκή πλευρά, διαφορετικά σίγουρα θα καταλήξουμε στα δικαστήρια. Νομίζω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το νέο κανονισμό προστασία των προσωπικών δεδομένων, το GDPR, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να στραφεί κατά των ΗΠΑ. Γιατί ουσιαστικά στην πράξη αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι παραβιάζεται και ένα άλλο σημαντικό κείμενο, ευρωπαϊκό και διεθνέ, το CRS, τα κοινά πρότυπα αναφορά. Στην πράξη δεν μπορεί να εφαρμοστεί ο ΦΑΤΚΑ, παρουσία του νέου αυτού κειμένου. Επίσης, ας μην ξεχνάμε ότι σε έκθεσή τους, οι φορολογικές αρχές των ΗΠΑ είπαν ότι μολονότι έχουν δαπανίσει εκατομμύρια ευρώ για τον ΦΑΤΚΑ, στην πράξη δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή την νομοθεσία. Ουσιαστικά καταστρέφουν τη ζωή αθώων Ευρωπαίων πολιτών που την χάνει να έχουν λόγω συγκυρία και την Αμερικανική υπηκότητα, χωρί να καταφέρουν καν οι αρχέ των ΗΠΑ να εισπράξουν τα χρήματα τα οποία θέλουν να εισπράξουν. Νομίζω ότι ε, γίνεται και μία παράλληλη συνεδρίαση σήμερα στις, στις Βρυξέλλες. Υπάρχουν εκπρόσωποι των γαλλικών αρχών. Υπάρχει και ο Μάρκος Νίτς από τις Ολλανδικές φορολογικές αρχές που είναι εδώ πέρα στις Βρυξέλλες και συμμετέχουν σε διαπραγματεύσεις για να καταφέρουν να προστατεύσουν τους Ολλανδούς υπηκόους που έχουν και την Αμερικανική υπηκότητα. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι ε, υπάρχει μια κάποια κινητοποίηση και από τη Βρετανική πλευρά. Υπάρχουν προφανώς Αμερικάνοι λόγω συγκυριών και, στις, ε, και στον Εμένο Βασίλειο. Και έπειτα έχουμε και την αποστολή αυτή της ε, γαλλικής κυβέρνησης που θα πάει στην Washington DC σύντομα. Τι γίνεται λοιπόν ακριβώ Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασία Δεδομένων δεν φαίνεται ότι μπορεί τελικά να τοποθετηθεί επισήμω επί του ΦΑΤΚΑ. Αυτό επιβεβαιώνει το πόρισμα του κυρίου Γκαμπαρίνο. Βλέπουμε ότι υπάρχουν ευρωπαϊκέ κυβερνήσει οι οποίε δεν θέλουν να μα δώσουν δεδομένα όσον αφορά τη ροή, τη ροή δεδομένων προ τι ΗΠΑ. Εμέσω παραδέχομαι ότι δεν υπάρχει καμία αμοιβαιότητα στη ροή των δεδομένων. τεράστιε ποσότητε δεδομένων πάνε στην Αμερική. ελάχιστε πληροφορίε έρχονται από την Αμερική προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από την άλλη βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλοί αρνητικές επιπτώσεις όσον αφορά και τον GDPR αλλά και την εφαρμογή των κοινών προτύπων αναφοράς. Διερωτάται λοιπόν κανείς για ποιο λόγο υπάρχει αυτή, για ποιο λόγο θελοτυφλούν ουσιαστικά οι ευρωπαϊκές αρχές. Νομίζω ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε καταβάλουν τεράστιε προσπάθειε για να εφαρμόσουν το ΦΑΤΚΑ. Του στοχίζει πάρα πολύ ακριβά αυτό. Ξέρω ότι το όλο ζήτημα στοιχίζει πάρα πολύ γενικότερα και στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Πάντω, οι τέσσερι μεγαλύτερε λογιστικέ εταιρείε όπω η PricewaterhouseCoopers, η KPMG κτλ. Έχουν, αρχίσει, έχουν σταματήσει μάλλον να κοινοποιούν στοιχεία όσον αφορά τον ΦΑΤΚΑ και όσον αφορά τον CRS βλέπουμε ότι στην πράξη δεν λειτουργεί το σύστημα αυτό. Είναι ένα σύστημα που έχουν επινοήσει οι Ηνωμένε Πολιτείε, από το οποίο δεν καταφέρουν να συγκεντρώσουν χρήματα και το οποίο στοιχίζει πάρα πολύ ακριβά στα ευρωπαϊκά τραπεζικά ιδρύματα. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εμεί ω Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τα κοινά πρότυπα αναφορά και πώς μπορούμε να ασκήσουμε πίεση στις Ηνωμένε Πολιτείε προκειμένου να επαναχωρήσουν τελικά και να σταματήσουν να ασκούν τέτοια πίεση στους Αμερικανούς πολίτες που διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του ΦΑΤΚΑ. Ναι, ναι, ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε. Δεν χρειάζομαι καν τα δύο λεπτά που μου δίνετε. Ουσιαστικά έχουμε μιλήσει με πάρα πολλούς αρμόδιους. Όλοι γνωρίζουν ότι οι Αμερικανοί λόγω συγκυριών υποφέρουν από τον ΦΑΤΚΑ. Έχουμε πάρα πολλούς εκπροσώπους και από την ευρωπαϊκή πλευρά και από την αμερικανική πλευρά. Κανείς δεν θέλει να κάνει τίποτα. Και οι Αμερικάνοι τι μας λένε. Εμεί δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή η οποία θα πρέπει να αρχίσει να προστατεύει ενδεχομένω του πολίτε τη. Μα λέει προφανώ ότι δεν είμαστε πλήρει Αμερικανικοί πολίτε. Αυτό ισχύει. Μπορεί να έχουν Αμερικανική υπηκότητα, δεν έχω ψηφίσει ποτέ στι ε, Ηνωμένε Πολιτείε. Επομένω, εναπόκειται στι ευρωπαϊκέ αρχέ να κάνουν κάτι, αλλά το θέμα είναι ότι νύπτουν τα χείρα του και οι ευρωπαϊκέ αρχέ. Αναφέρονται σε διάφορε διεθνεί συμφωνίε, οι οποίε ισχύουν και ουσιαστικά προσπαθούν να αποφύγουν, αν θέλετε, να αντιμετωπίσουν το ζήτημα αυτό. Θέτω λοιπόν το εξή ρητορικό ερώτημα. Αν είχατε ένα παιδί και το παιδί αυτό είχε δύο γονιού και ένα από του γονεί αυτού κακοποιούσε το παιδί, ο άλλο γονιό τι, θα έπρεπε, τι θα έπρεπε να κάνει. Θα έπρεπε ουσιαστικά να κάθεται με τα χέρια σταυρωμένα και να μην κάνει τίποτα, λέγοντα ότι ουσιαστικά ο γονιό ο οποίο κακοποιεί το παιδί του έχει και το προνόμιο να κάνει κάτι τέτοιο, ότι αυτό προβλέπεται στα πλαίσια τη γονική μέρημνα, ή θα έπρεπε άλλο γονιό να αναλάβει δράση και να σταματήσει αυτή η παράνομη δράση. Αυτό ακριβώ νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε και προκειμένου. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η αναφορά αυτή και η απάντησή μας, όπως ε, εξήγησε ο αναφέρον, έχει να κάνει με τρία θέματα. Η ιδιωτική ζωή, προστασία δεδομένων, δηλαδή πιθανή διάκριση στις ευρωπαϊκές ε, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ε, σύμφωνα με την οδηγία περί πληρωμών, καθώς και τον νόμο ΦΑΤΚΑ αυτών καθ' που έχει κάποιες φορολογικές συνέπειες λόγω του ορισμού του φορολογούμενου από πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει απαντήσει επισήμω στα θέματα αυτά. Επειδή το θέμα αυτό αφορά τρία, τρεις, τρία τμήματα της Κομισιόν, εγώ θα μιλήσω για το φορολογικό θέμα, ενώ οι συνάδελφοί μου θα επανέλθουν ε, όσον αφορά ε, την προστασία των δεδομένων και την εφαρμογή του ε, κανονισμού της οδηγίας περιπληρωμών. Έχουμε λοιπόν 28 κράτη-μέλη τα οποία συμφώνησαν με τις Ηνωμένε να ανταλλάσσουν πληροφορίες. Οι πληροφορίες που παρέχουν ε, είναι πολύ παρόμοιες ε, με αυτές που έχουν συμφωνήσει και άλλα κράτη να υποβάλουν σύμφωνα με το κοινωνικό σύστημα υποβολής ε, στοιχείων. Και εντό Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε την οδηγία για τη διοικητική συνεργασία. Οι πληροφορίε αυτέ λοιπόν που ανταλλάσσονται είναι λίγο πολύ ίδιε. Υπάρχει λιγότερη αμοιβαιότητα με τι ΗΠΑ, διότι οι ΗΠΑ δεν φαίνεται να παρέχουν τι ε, εξίσου πολλέ πληροφορίε στα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, δεν έχουμε πρόσβαση εμεί στα δεδομένα αυτά. Είναι εθνικέ συμφωνίε που έχουν συμφωνήσει τα κράτη-μέλη σε απάντηση της επιθυμίας του Κοινοβουλίου για αναθεώρηση της ΦΑΤΚΑ είπαμε ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε με τις πληροφορίες που έχουμε στα χέρια μας. Είμαστε διατεθειμένοι να, να συζητήσουμε με το Συμβούλιο και αν το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη θέλουν να μας δώσουν εντολή θα τη δεχτούμε για να συζητήσουμε με τις ΗΠΑ πώς μπορεί ο ΦΑΤΚΑ να εφαρμόζεται με πιο σωστό τρόπο σε ανθρώπους με διπλή υπηκότητα. Το θέμα είναι ακριβώς οι άνθρωποι με διπλή υπηκότητα, διότι οι οι Ηνωμένε Πολιτείε φορολογούν τους πολίτε, τους υπηκόου των Ηνωμένων Πολιτείων, ενώ οι άλλε χώρε του κόσμου ε, φορολογούν του ε, διαμένοντες, τους κατοίκου τη χώρα τους. Είπαμε λοιπόν ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά κάτι που μπορώ να προσθέσω είναι ότι ο Επίτροπός μας, ο κύριος Μοσκοβίση, έχει συζητήσει με τις Ηνωμένε Πολιτείες σε το θέμα αυτό του ΦΑΤΚΑ και συζητήθηκε το πώς μπορεί να γίνει πιο εύκολο για τους ανθρώπους με διπλή υπηκότητα να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους. Ε, φαίνεται λοιπόν να υπάρχουν εξελίξεις, ε, είναι όμως ακόμα σε άτυπο επίπεδο. Όσον αφορά το να γίνει πιο εύκολο να απαλλαγεί κανείς από την υπηκότητα, αυτό δεν έχει ε, συζητηθεί ακόμη, ούτε ε, έχουν γίνει προσπάθειες να πείσουμε τις Ηνωμένε Πολιτείες να ε, αλλάξουν πολιτική όσον αφορά την, την φορολογία. Αυτά όσον αφορά τη φορολογία, αλλά θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους μου για τα θέματα προστασίας δεδομένων και πληρωμών. Καλή σας μέρα. Νικολό Μπρινιόλη ε, από την Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες ε, και μιλώ ιδιαίτερα για την ε, οδηγία περί πληρωμών. Ε, ακούσατε αυτά που είπε ο συνάδελφός μου όσον αφορά το θέμα της φορολογίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με το πώς οι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζουν δυσκολίες ε, λόγω του νόμου ΦΑΤΚΑ. Ο χρηματοοικονομικός ε, τομέας έχει επισημάνει επανειλημμένα ότι ε, ο αριθμός ε, ταυτότητας ε, για την ΦΑΤΚΑ έχει δημιουργήσει προβλήματα. Τον Μάρτιο του 2017 ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Αρμόδια Αρχή να εξετάσει πόσοι οι υπήκοοι και πόσες τράπεζες δεν μπόρεσαν να ανοίξουν λογαριασμό πληρωμών. Μία εθνική αρχή μόνο είχε λάβει επίσημη προσφυγή όσον αφορά το ΦΑΤΚΑ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης έθιξε το θέμα αυτό με διακρατική ομάδα επιρροχνωμόνων τον Απρίλιο του 2018 και έλαβε παρόμοια ανταπόκριση από πλευρά των κρατών μελών. Σύμφωνα με την Οδηγία περί λογαριασμών πληρωμών, όλοι οι κάτοικοι που κατοικούν ε, νόμιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των κατατύχει Αμερικανών και των πραγματικών Αμερικανών, ε, έχουν δικαίωμα να ανοίξουν ε, έναν τέτοιο λογαριασμό τα κράτη-μέλη είναι αρμόδια για την εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας που ε, εφαρμόζει την ε, οδηγία όσον αφορά το συγκεκριμένο δικαίωμα. Σε συνέχεια ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πέρυσι το καλοκαίρι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διενεργήσει ανάλυση της μεταφοράς στο Εθνικό Δίκαιο των σχετικών άρθρων ε, της οδηγίας, ιδιαίτερα το άρθρο 15 για μη διάκριση και το 16 για ε, το δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα κράτη-μέλη και τα 28. Δεν μπόρεσε όμως ε, να διαπιστώσει συγκεκριμένα προβλήματα όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ελισαβέκεμαν από τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης. Ακούσαμε κάποια θέματα στην παρουσίαση. Ακούσαμε και τον καθηγητή Καπαρίνο που μίλησε εδώ πέρσι. Ε, στην έκθεσή του ε, έλεγε ότι δεν ε, ισχύουν πια τα περί προστασίας δεδομένων, διότι τα άτομα δεν θα έχουν πια δικαίωμα προσφυγή σε σύμφωνα με ε, τον κανονισμό για την προστασία των δεδομένων. Ε, δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο για συμμόρφωση με το, την ομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των δεδομένων. Υπάρχουν συμφωνίες ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένε Πολιτείες. Έχουμε ε, και την σύμβαση του ΟΣΑ που λέει ότι τίποτα στην ε, σύμβαση αυτή δεν θίγει δικαιώματα που ε, προκύπτουν από την εθνική νομοθεσία. Και οι αρχές λοιπόν και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν διαφάνεια και να απαντούν σε αιτήματα υποκειμένων των δεδομένων. Υπάρχουν κάποιε συγκεκριμένε υποχρεώσει ε, όσον αφορά την προστασία δεδομένων από πλευρά ε, των χρηματοπιστωτικών ε, οργανισμών και των αρχών. Κάθε άτομο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να υποβάλει προσφυγή όσον αφορά την προστασία δεδομένων στο πλαίσιο της ΦΑΤΚΑ στην αρχή προστασίας δεδομένων. Έχει επίσης πρόσβαση στα εθνικά δικαστήρια για τα θέματα αυτά. Στο πλαίσιο του ΦΑΤΚΑ, λοιπόν, ε, θα χρειαστεί ε, συγκεκριμένη εξέταση κατά περίπτωση ε, αν υπάρχει πρόβλημα. Οι ανεξάρτητες εθνικές αρχές όμως είναι καλύτερα σε θέση να αξιολογήσουν την κατάσταση. Και το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων έχει αποφανθεί σχετικά με τον ΦΑΤΚΑ στο παρελθόν, για παράδειγμα πέρσι τον Μάιο, είπαν ότι δεν διαπιστώθηκε ε, ότι θα πρέπει να απαγορευτούν οι οι ε, μεταφορές ε, στοιχείων σύμφωνα με τον ΦΑΤΚΑ. Εξετάστε το θέμα αυτό πιο αναλυτικά για να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση στα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετέχει στο Συμβούλιο για την Προστασία των Δεδομένων και παρακολουθούμε στενά τι εξελίξει στο θέμα αυτό. Σα ευχαριστώ. Χρόνο για του συναδέλφου κυρία Σόφη Ιντβέλτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι απογοητευτικό να ξανασυζητάμε αυτό το θέμα. Πάλι. Ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων ε, στους εκπροσώπους Κομισιόν, γιατί οτιδήποτε που δεν τους αφορά προσεκτικά, διακρίνω αφενός την πολιτική ως πολιτικό σώμα που είναι υπεύθυνο ή θα έπρεπε να είναι υπεύθυνο, και εσά που είσαστε απλοί άνθρωποι που κάνετε τη δουλειά σας. Ειλικρινά όμω σας λέω, είναι προφανέστατο ότι η Κομισιόν, το πολιτικό σώμα, επιλέγει να μην αντιμετωπίσει αυτό το θέμα. Μα Γιατί σε πολλούς τομεί η, ε, η Κομισιόν ε, είναι το, το σκυλάκι τον ύπα. Αν οποιαδήποτε άλλη χώρα ε, ενοχλούσε τους πολίτες, ευρωπαίους πολίτες με διπλή ε, ηθαγένεια με αυτόν τον τρόπο, θα, θα υπήρχαν ακόμα αμέσως δηλώσεις από τη Μογκερίνη και τον Γιούγκερ κτλ. Με τους Αμερικανούς, α, ξαφνικά είσαστε, γινόσαστε επιθύμια όργανα. Έχετε, παραδείγματο χάρη, αρμοδιότητα για να κάνετε δηλώσεις αντίον της Τουρκίας. Όχι, αλλά δεν σας εμπόδισε, ας πούμε, για να κάνετε δηλώσει και να στείλετε και 6 δισεκατομμύρια στην Τουρκία. Γιατί λοιπόν ξαφνικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει τι ευθύνε τη, Συγγνώμη, αλλά για να σας ακούω ο, να το αντιμετωπίζετε τόσο γραφειοκρατικά το θέμα αυτό, πραγματικά με βάση την οδηγία ας πούμε, για τους λογαριασμούς πληρωμών και να μας λέτε στο τέλος ότι κάναμε μια σοβαρή εξέταση, εξετάσαμε το τάδε κουτάκι, το δίνα κουτάκι κτλ. και δεν υπάρχει πρόβλημα. Μα είναι άνθρωποι αυτοί οι συγκυριακοί Αμερικανοί. Έχουν ε, σάρκα και οστά, μπορείτε να τους αγγίξετε. Υπάρχουν πάρα πολλά δεδομένα ε, από αυτούς τους ανθρώπους, μα μας γράφουν αυτοί οι άνθρωποι, ξέρουμε ότι υπάρχουν. Γιατί εσείς εθελοτυφλείτε, κάνετε σαν μην υπάρχουν. Είναι εντυπωσιακό. Αυτό έχει να κάνει με το πώς ε, αντιμετωπίζετε τις είπα, Πριν από τα Χριστούγεννα, μπορεί να το διάψουν στον τύπο, χωρί να ενημερωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένε Πολιτείε αποφάσισαν να υποβαθμίσουν το διπλωματικό καθεστώ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι μα αντιμετωπίζουν. Σαν δούλου. Εσεί θα πρέπει να ορθώσετε το ανάστημά σα και να υπερασπιστείτε τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Ε, υποτίθεται ότι η Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια σημαίνει κάτι, το να είσαι Ευρωπαίο πολίτη. Υποτίθεται ότι κάτι σημαίνει. Νομίζω ότι οι κατατύχοι αυτοί οι Αμερικανοί είναι τα θύματα τα οποία πραγματικά ε, είναι... Θυματοποιήθηκαν ε, γιατί στην πραγματικότητα είναι στη μέση, βρέθηκαν στη μέση. Εσείς τι λέτε τώρα, μας ενδιαφέρουν αυτοί οι άνθρωποι. Εκλογικά μετράνε, Όχι. Μπα, δεν θα κάνουμε τίποτα. Το ξεχνάμε. Κάτω από το χαλί το, το στέλνουμε. Τι πρέπει να κάνουμε, κατά τη γνώμη μου, Θα πρέπει να οργανώσουμε μια σύνοδο όπου καλούμε. Θα καλέσουμε το Μοσκοβισί και ε, από χώρες ε, πολιτικούς από την Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, από ε, χώρες όπου κάτι κινείται και να το συζητήσουμε πριν τις εκλογές. Γιατί δυστυχώς μετά το καλοκαίρι τίποτα δεν θα κάνει, θα περιμένουν όλη τη νέα Κομισιόν και το νέο Κοινοβούλιο. Μετά τι εκλογέ δεν θα γίνει τίποτα λοιπόν. Α κάνουμε ένα κύκλο, ένα, μια συζήτηση στρογγυλή τραπέζη πριν τι εκλογέ, ούτω ώστε να έχουμε μια κοινή στρατηγική για αυτού του ανθρώπου και να αναλάβουμε, εν πάση περιπτώσει, τις ευθύνες μας και να αναλάβει και η Κομισιόν τις ευθύνες της. Δεύτερον, η Κομισιόν και ίσως η Επιτροπή Αναφορών να ζητήσει ε, επίσημα από την ε, Κομισιόν να υπάρχει ένα γραφείο όπου τα θύματα του ΦΑΤΚΑ να πηγαίνουν κατευθείαν και να αναφέρουν το πρόβλημά τους, ούτως ώστε να μην λέει η Κομισιόν πια και να μην ισχυρίζεται ότι «Α, εγώ δεν έχω ιδέα ποιο έχει δυσκολίε. θα πρέπει κάπου να βρεθεί ένας υπάλληλο που έχει χρόνο για να διεκπεραιώνει τα παράπονα των θυμάτων του ΦΑΤΚΑ, ούτω ώστε να έχουμε μία εικόνα για την κλίμακα του προβλήματος. Αυτές είναι οι δύο προτάσεις που σας υποβάλλω. Κύριε Ροζιέρ, σας ευχαριστώ. Συμφωνώ απόλυτα με την Σοφή Ινβέλτ. Ειλικρινά, δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά πόσες φορές ακόμα σε αυτό το ζήτημα αλλά και σε άλλα θα βλέπουμε Ευρωπαίους πολίτες των οποίων τα δικαιώματα παραβιάζονται, τα δικαιώματα των οποίων υποτίθεται ότι εμεί πρέπει να προστατεύουμε, και έρχονται εδώ πέρα και μα λένε ότι καταπατώ τα δικαιώματά του και η μόνη απάντηση που λαμβάνουν είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, δεν είναι δική μα αρμοδιότητα, το εξετάσαμε το ζήτημα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και ειλικρινά αυτή τη στιγμή δεν στρέφουμε προσωπικά κατά των εκπροσώπων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχουμε εδώ σήμερα και ξέρω ότι και το δικό του το έργο είναι δύσκολο γιατί το δικό του το θεσμικό όργανο του αναγκάζει να είναι εκπρόσωποι τελικά να εκπροσωπούν τη βία αυτή απέναντι στους πολίτες αυτής. Και ουσιαστικά στους πολίτε αυτού τι λέμε, δεν υπάρχετε, δεν υφίσταστε και δεν υπάρχουν καν τα δικαιώματά σα και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για σας και δεν ενδιαφερόμαστε καθόλου. Και μετά ακούμε όλα αυτά τα μεγαλεπίβολα λόγια, για ποιο λόγο άραγε οι Ευρωπαίοι πολίτε ε, δεν ε, έχουν εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για ποιο λόγο δεν συντάσσονται με το ευρωπαϊκό σχέδιο, με το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, για ποιο λόγο δεν καταφέρουμε να τους πείσουμε ότι είμαστε αξιόπιστοι και το καθεξής. Ε, μα ορίστε, να η απόδειξη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να συζητάμε τέτοια ζητήματα, να πηγαίνουμε μετά και να εξηγούμε την νομοποίηση που μας δίδεται, το ρόλο που υποτίθεται ότι επιτελούμε εδώ πέρα, την αποτελεσματικότητα που υποτίθεται θα έπρεπε να έχουμε. Πραγματικά δεν ξέρω αποτιμάτε τη βία την οποία υφίστανται αυτοί οι άνθρωποι. Άνθρωποι οι οποίοι στρέφονται προς εμάς, μας λένε εσείς μας εκπροσωπείτε, εσείς είστε η εκτελεστική δύναμη, εσείς υποτίθεται ότι θα πρέπει να προσπίσετε τα δικαιώματά μου και η μόνη απάντηση που λαμβαίνουν είναι α, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και μάλιστα ακόμα χειρότερο. Δεν είμαστε καν σίγουροι ότι υπάρχει πρόβλημα, αυτό τους λέμε. Πραγματικά είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα και ειλικρινά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να δείχνουμε ε, τέτοια διαφορία απέναντι στους πολίτες και έχει απόλυτο δίκιο η Σοφίντ Βέλτε. Ενδεχομένως θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άμεσος διάβλος ανάμεσα στους πολίτες και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ενδεχομένως με τις άμεσες αυτές επαφές ε, θα συνειδητοποιήσουν ορισμένοι ότι το πρόβλημα υφίσταται πραγματικά και ότι κάτι πρέπει να γίνει γι' αυτό. Και βέβαια δεν εμπλέκεται μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και εθνικέ κυβερνήσει. Και το πρόβλημα είναι ότι ο ένα στέλνει τον μπαλάκι στον άλλον, κανεί δεν αναλαμβάνει ευθύνη, δεν είναι δική μου αρμοδιότητα, φταίνει οι υπόλοιποι και το καθεξής. Αυτά ακούν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Και νομίζω ότι έχετε απόλυτο δίκιο πραγματικά. Κάθε φορά που βλέπουμε ότι διακυβεύονται οικονομικά συμφέροντα ουσιαστικά που πονάνε, τότε ξαφνικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανασυντάσσεται και βρίσκει τρόπους για να ασκήσει πίεση και το καθεξής. Εκεί πέρα πραγματικά καταφέρνουμε και καταγγέλουμε διάφορα κακό κείμενα. Ε, μήπως θα έπρεπε και προκειμένου να κάνουμε κάτι τέτοιο. Μήπως θα έπρεπε να ανασυνταχθούμε και για το ζήτημα αυτό. Πολύ σύντομα θα ε, λήξει το μορατόριο αυτό των ΗΠΑ. Ενδεχομένω λοιπόν θα πρέπει υπεύθυνοι, μη τι άλλο, να ανασυνταχθούν, να κινηθούν και μέχρι τα τέλη του έτου να καταφέρουν να βρουν μια λύση. Το μορατόριο αυτό το οποίο ουσιαστικά επιτρέπει στις τράπεζες να μην υποβάλουν ακόμα τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης, τον αριθμό φορολογικού μητρώου των πολιτών. Αλλά καταλαβαίνετε ότι η προθεσμία αυτή θα εκπνεύσει στα τέλη του έτους και θα αναγκαστούν και τα δεδομένα αυτά να διαβιβάζονται προς τις Ηνωμένε Πολιτείε. Ίσως λοιπόν να πρέπει όντως τώρα να κινητοποιηθείτε. Εμεί σε κάθε περίπτωση με την Τζουντ, με τη Σοφή και με όλου του ενδιαφερόμενους συναδέλφου θα συνεχίσουμε να καταβάλουμε προσπάθειες γιατί θεωρούμε ότι είμαστε πραγματικά οι εκπρόσωποι των ανθρώπων αυτών οι οποίοι, των οποίων μάλλον τα δικαιώματα καταπατώνται και εναντίον των οποίων υφίστανται αυτή τη στιγμή πολλές μορφές διακριτικής μεταχείρισης. Νομίζω ότι δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να κλείσουμε με τέτοια αναφορά. Τα προβλήματα αυτά βρίσκονται σε εξέλιξη και συνεχίζονται. Οφείλουμε λοιπόν να κρατήσουμε ζωντανή την αναφορά αυτή και σίγουρα είναι απογοητευτικό και για μας αυτό, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε να εκπροσωπούμε τους πολίτες αυτούς, γιατί αυτός άλλωστε είναι και ο ρόλος μας που έχουμε ω ευρωβουλευτέ. Πρέπει να συνεχίσουμε να του υπερασπιζόμαστε. Σα ευχαριστώ πολύ, κυρία Κέρτσον Ντάρλινγκ. Συμφωνώ με πολλά από όσα υπόθηκαν. Πιο πολύ νιώθω το εξής. Είναι κατανοητό το γιατί είναι τόσο οργισμένοι οι άνθρωποι, αυτοί οι accidental Americans, οι κατατύχοι Αμερικανοί. Είναι κατανοητό το ότι είναι οργισμένοι από την αδράνεια των αρχών που υποτίθεται ότι προστατεύουν τα δικαιώματά τους σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως θεσμικό όργανο, θα πρέπει να στραφούμε, όχι ε, ε, κατά εσάς προσωπικά, αλλά κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, διότι είχαμε εξηγήσει σαφώς τι θα θέλαμε να δούμε ως ευρωπαϊκή αντίδραση, συντονισμένη δράση, μία σαφή στρατηγική. Και από ό,τι καταλαβαίνω, Ε, ο συντονισμός ε, μέχρι τώρα δεν φαίνεται να πηγαίνει πολύ καλά. Έχουμε τρεις ανθρώπους από τρεις διαφορετικές υπηρεσίες τη επιτροπή που μας ε, μιλάνε εδώ. Δεν βλέπω να υπάρχει συντονισμένη στρατηγική όσον αφορά τον νόμο ΦΑΤΚΑ και τις συνέπειες για τους κατατύχει Αμερικανού. Και νομίζω ότι αυτό είναι προσβολή και απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. έχει υιοθετηθεί ψήφισμα με ουσιαστικά τεράστια πλειοψηφία στο πλαίσιο της ε, πολιτικής δυναμικής του Κοινοβουλίου πρόκειται για πραγματικά μεγάλη πλειοψηφία. Θίγει λοιπόν ε, το Κοινοβούλιο το θέμα αυτό και συμφωνώ με τη Σόφη ότι είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Εγώ γεννήθηκα στην Τανζανία, έφτασα στο Ηνωμένο Βασίλειο όταν ήμουν 11 μηνών και ούτε δεν μπορώ να φανταστώ ποια θα ήταν η αντίδραση εάν η Τανζανία άρχιζε να φορολογεί το μισθό μου. Αμερικανοί που έχουν γεννηθεί στις Ηνωμένε Πολιτείε, κατά τύχη Αμερικανοί δηλαδή, γεννήθηκαν στις Ηνωμένε Πολιτείε, επέστρεψαν στην Ευρώπη σε ηλικία 11 μηνών και τώρα ε, δέχονται αυτό το δρακόνιο σύστημα. Είναι λοιπόν θέμα πολιτικής βούλησης και ο ρόλος μας ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι να υπερασπιστούμε τους ε, ανθρώπους αυτούς και να μην ε, σκουπίσουμε τη σκόνη κάτω από το χαλί. Και να αφήσουμε το θέμα αυτό εκρεμές σε αυτήν την ε, την ε, συγκεκριμένη χρονική στιγμή όπου έχουμε ευρωεκλογέ, ε, οπότε όλα θα μείνουν κάπως στον αέρα. Συμφωνώ λοιπόν ότι θα πρέπει να κινηθούμε όσο γίνεται πιο γρήγορα πριν τις εκλογές. Και αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό για τους Βρετανούς κατά τύχη Αμερικανούς, ε, διότι ο ε, αναφέρον ήταν αρκετά μεγαλόψυχος απέναντι στο Ηνωμένο Βασίλειο στην παρουσίασή του. Είναι θλιβερό το πόσο καιρό έχει αγνοηθεί το θέμα τελείως ε, στο Westminster. Εγώ το έχω θίξει αυτό με τους αρμόδιες ε, της πολιτικής μου ομάδας, αλλά δεν νομίζω ότι ούτε αυτοί έχουν ε, λάβει υπόψη του σοβαρά το θέμα. Έχουμε κάποιους εξαιρετικούς βουλευτές που αγωνίζονται για το θέμα αυτό ε, υπερασπίζοντας τους ψηφοφόρους τους, ε, αλλά πρόκειται για μια πολύ μικρή ομάδα. Και μόνο λόγω της πίεσής τους ο ε, Μέλστραιντ έχει αρχίσει να απαντάει ως αρμόδιος υπουργός. Εμένα λοιπόν η ανησυχία μου είναι ότι με το Brexit για τους Βρετανούς κατά τύχη Αμερικανούς όταν βρεθούμε πάλι στις ανοιχτές θάλασσες της παγκόσμιας πολιτικής, ξέρουμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ε, ε, απελπισμένα προσπαθεί να μην ε, προσβάλλει τις Ηνωμένε Πολιτείε. Η εξολόγηση μου είναι λοιπόν ότι θα δυσκολέψει ακόμη πιο πολύ η κατάσταση για τους Βρετανούς ε, κατά τύχη Αμερικανούς και θεωρώ ότι έχω ηθική ευθύνη να διατηρήσουμε την αλληλεγγύη αυτή που υπάρχει ανάμεσα στους κατήχοι Αμερικανούς στην Ευρώπη, ασχέτως από το σε ποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμένουν. Αλλά φαντάζομαι ότι από οργανωτικής πλευράς θα είναι εφιάλτη στο να οργανωθεί οτιδήποτε εντός του Κοινοβουλίου από τώρα μέχρι τις ευρωεκλογέ. Σας καλώ όμως να σκεφτούμε ε, με καινοτόμο τρόπο να ε, επιστρατεύσουμε την φαντασία μας για να βρούμε καλή λύση και να προσπαθήσουμε ως Κοινοβούλιο να ζητήσουμε λογοδοσία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με το ψήφισμα που υιοθετήσαμε τον Ιούλιο. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι όλοι είχαν τη δυνατότητα να πάρουν το λόγο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συζήτηση αυτή. Έχουμε μια πρώτη αντίδραση από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γραπτός. Έχουμε και τη γνωμοδότηση των Επιτροπών ΕΚΟΝ και ΛΥΜΠΕ. Είχαμε μια αρκετά ολοκληρωμένη συζήτηση στο Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό. Και θα ήθελα να πω το εξής, το οποίο θεωρώ ότι είναι σωστό. Ακούστηκαν πολλές επικρίσεις κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συμφωνώ με τις επικρίσεις, αλλά δεν θα πρέπει αυτή η κριτική να στρέφεται κατά των εκπροσώπων της Κομισιόν που είναι παρόντες, ε, θα πρέπει να στρέφεται κατά του πολιτικού επίπεδου. Και για το λόγο αυτό προτείνω να κάνουμε το εξή. Η αναφορά αυτή φυσικά θα παραμείνει ανοιχτή. Δεύτερον, Έχουμε ξανασυζητήσει το θέμα αυτό και προτείνω το ίδιο που πρότεινα και την προηγούμενη φορά. Να στείλουμε μία σαφή επιστολή στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών για να επισημάνουμε το θέμα αυτό στις Αμερικανικές αρχές και επίσης προτείνω να στείλουμε επιστολή στον Επίτροπο Μοσκοβισή, ενδεχομένως με αντίγραφο προς τον κύριο Γιούγκερ. Διότι και οι τρεις εκπρόσωποι της Κομισιόν είπαν ότι πιστεύουν ότι υπάρχουν δυνατότητες, χρειάζεται όμως πολιτική απόφαση υψηλό επίπεδο. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα χρονοδιάγραμμα από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τέταρτον, Νομίζω ότι θα πρέπει να συμμετέχουν και τα κράτη-μέλη. Προτείνω λοιπόν να στείλουμε επιστολή προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, καλώντας τον ε, να ε, στραφεί στα κράτη-μέλη, τα κράτη-μέλη να αξιολογήσουν την κατάσταση και να ε, πούν πώς πιστεύουν ότι μπορούμε να προχωρήσουμε. Αρκούν αυτά. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν, κάθε επιτυχία σας εύχομαι και ολοκληρώνουμε έτσι το θέμα αυτό. Και φτάνουμε στην αναφορά 252 του 2018 ε, από τη Σλοβακία. Πρόκειται για την αναφορά της Ρενάτα Παπκούνοβα. Παπτσούνοβα και έχει να κάνει με την δολοφονία του Σλοβάκου δημοσιογράφου Γιάν Κούτσιακ. Και της αραβωνιαστικιάς του Μαρτίνα Κουσνίροβα. Περνάμε λοιπόν σε αυτό το θέμα της ημερησίας διάταξης. Καλωσορίζω την αναφέρουσα, την ε, κυρία Παψούνοβα. Έχετε το λόγο. Η ελευθερία, η ασφάλεια και η δικαιοσύνη είναι ο στόχος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακριβώς γι' αυτό τόσο πολλοί άνθρωποι υπέγραψαν αυτή την αναφορά. Πάνω από 60.000 άνθρωποι πιστεύουν ότι δεν υπάρχει ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη στη Σλοβακία. Είμαι ενώπιόν σας. Εδώ δεν είμαι... Α, είμαι ακτιβίστρια, δεν είμαι δημοσιογράφος, δεν είμαι πολιτικός, δεν έχω σκοπό να γίνω πολιτικός. Ε, δουλεύω για μία ΜΚΟ. Είμαι μητέρα, εργαζόμενη και Σλοβάκα. Και θέλω να σας πω τι συμβαίνει στη χώρα μου και στη δημοκρατία της. Το περασμένο Σάββατο, 9 από τους 13 συνταγματικούς δικαστές ε, ολοκληρώσαν τη 12η θητεία τους ε, και το Κοινοβούλιο όμως δεν εξέλιξε τους καινούριου, γιατί το, το 45% των μελών αποφάσισαν να μην ε, ρίξουν έγκυρη ψήφο. Είχαν δύο ευκαιρίες σε δύο μέρες αλλά παρόλα αυτά αποφάσισαν να αγνοήσουν το δικαστικό μας σύστημα, γι' αυτό το σύστημά μας βρίσκεται σε φοβερή κρίση. Πριν λίγες μέρες μάθαμε κάτι για αυτόν τον άντρα, τον Τουσάν Κόβατσικ, έναν ειδικό εισαγγελέα που κατηγορήθηκε για πολλά σοβαρά οικονομικά εγκλήματα στη Σλοβακία. Το 2017 έφερε στην τράπεζα πάνω από 200.000 ευρώ σε ρευστό και τα έβαλε στο λογαριασμό του. Η τράπεζε το ανέφεραν, αλλά η αστυνομία το αγνόησε. Αυτό ο άνθρωπο ήταν επικεφαλή για 61 σοβαρά οικονομικά εγκλήματα κατά τα 8 χρόνια που ήταν στο θόκο τον δικαστικό, αλλά κανένας δεν δικάστηκε από αυτούς. Προχωρώ. Ε, η Υπουργό Εσωτερικών, Τενίσα Σάκοβα, την περασμένη εβδομάδα, η Υπουργό αυτό αποφάσισε ορισμένες από τις έρευνες να τις ε, αφαιρέσει από την αστυνομία και να τις αναλάβει αυτή. Και ο κύριος Λίψικ και ο κύριος Κβάστινα, ε, οι δικηγόροι που εκπροσωπούσαν τον Γιάννη και την Μαρτίνα και τις οικογένειές τους, ε, διαφώνησαν και είπαν ότι η αστυνομία δεν είχε τους πόρους ή την αρμοδιότητα να ασχοληθεί με έρευνες για δολοφονία. Η Υπουργό Σάκοβα είπε ότι αποφάσισε αυτό που αποφάσισε μαζί με τον πρώην πρόεδρο της αστυνομίας Τίμπορ Γκάσπα. Αυτός, ο Τίμπορ Γκάσπα, είναι αυτός ο οποίος ε, παρετήθηκε γιατί τον πίεσε ο λαός. Ε, ο κόσμος είπε ότι δεν έχει εμπιστοσύνη στην εξαρτησία του. Ε, είπε ψέματα ε, στην αρχή της έρευνας και έχει σχέσεις με τον ολιγάρχη Μπόντορ που πήρε ε, εκατομμύρια από το κράτος και από ευρωπαϊκά κονδύλια. Ε, και ο δημοσιογράφο αυτό που σκοτώθηκε έγραψε για αυτόν. Ένα άλλο φοβερό γεγονό που μάθαμε την περασμένη εβδομάδα είναι ο κ. Μποροβτζόφ, που είναι επικεφαλή ε, τη Υπηρεσία Πληροφοριών τη ε, Οικονομική Αστυνομία, ε, παραδέχτηκε ότι έλεγξε τον λογαριασμό, τον φάκελο του Ιαν κατόπιν εντολή του τότε επικεφαλή αστυνομία Τίμπορ Γκάσπαρ. Αυτό έγινε το φθινόπωρο του 2017, μήνε πριν δολοφονηθεί ο Γιάννη και η Μαρτίνα. Ε, εκείνη τη στιγμή ε, ο δημοσιογράφος ε, ανέφερε ότι απειλήθηκε, αλλά τον αγνόησαν. Ο Τίμπορ Γκάσπαρ πήγε από τη θέση του ως επικεφαλής αστυνομίας στο, Υπουργείο Εσωτερικών ως σύμβουλος. Κάτι άλλο πρόσφατο. Ο Ζόλντοαν Αντρούσκο παραδέχτηκε ότι υπήρχε σχέδιο να δολοφονηθεί ο πρώην Υπουργό ε, Δικαιοσύνη, Ντάνιελ Λίψικ, που αυτή τη στιγμή εκπροσωπεί ω δικηγόρο την οικογένεια του Γιάνν Κούτσιακ. Και υπήρχε, ε, ήταν επικηρυγμένο για να τον δολοφονήσουν και θα δίνανε στο δολοφόνο του 200.000 ευρώ. Α, παραδέχτηκε επίση, ότι είχε ε, σχέδιο να σκοτώσουν και τον Γιάνν ε, που είναι ε, αναπληρωτής γενικού εισαγγελέα ε, αναπληρωτής ε, γενικός, ε, Ε, δεν μπορώ όμως να κάνω αυτή την παρουσίαση χωρί να αναφέρω ε, το πιο, τους πιο ισχυρούς άντρες στη Σλοβακία που αδιαφορούν για την ε, ασφάλεια του έθνους μας. Ο Ρόμπερτ Φίκο, πρώην ε, Πρωθυπουργό και αρχηγός του μεγαλύτερου κόμματος και ο σύμβουλός του που είναι γυναίκα, η κυρία Τρόσκοβα. Η κυρία Τρόσκοβα είχε σχέσεις με τον κύριο Βάνταλα, με Ιταλικέ επιχειρήσει ε, και επιχειρηματίε που ζούσαν στη Σλοβακία και σχέση με την ιταλική μαφία ε, και υπάρχει και ένταλμα σύλληψη στην Ιταλία εναντίον του, του κ. Βάνταλα. Επίση, πήρε πάρα πολλά λεφτά από ευρωπαϊκά κονδύλια, από αγιορικέ δραστηριότητε κτλ. Και ο κ. Γιάνν Κούσιακ έγραψε για αυτόν τον κύριο, ε, για τον κύριο Βάνταλα και τη σχέση με την Ιταλία και τη μαφία. Ε, η κυρία Τρόσκοβα ε, επίση ε, ήταν παρούσα σε πολλέ ε, επίσημε επισκέψει του Ρόμπερτ Φίκο ε, και όταν επισκέφτηκε την ε, καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ. Δεν ξέρουμε πολλά πράγματα. Ο κύριος Κάλινακ, ε, πρώην Υπουργό Εσωτερικών, υποτίθεται ότι εμπλέκεται στην απαγωγή ενός Βιετναμέζου επιχειρηματία, ο οποίος ζητούσε άσυλο στη Γερμανία, τον φέρανε στη Σλοβακία και τον έστειλαν με πτήση στο, στην ε, Μόσχα, όπου ε, τον δίκασαν και του έδωσαν, ε, τον καταδίκασαν ε, σε ισόβια. Ο κύριος Κάλινακ ε, είπε ότι δεν έχει καμία σχέση με την απαγωγή αυτή, όμως υπήρχαν ασυμβατότητες ανάμεσα στη ιστορία που είπε. Ε, επίσης, η επίσημη επίσκεψη που είχε, γίνει, ε, που είχε κάνει ε, στο Βιετνάμ ε, οργανώθηκε τελευταία στιγμή, ας πούμε. Επίσης, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Αντρέι Ντάνκο, που υποθέτει κάνει δοκτορά Πρόσφατα η Επιτροπή του Σλοβακικού Πανεπιστημίου επιβεβαίωσε ότι αντέγραψε 63 από τις 72 σελίδες από, την, από το δακτορικό του και δεν ζήτησε ούτε συγγνώμη. Και έπειτα έχουμε τον Υπουργό ε, ο οποίος ενέκρινε 33 εκατομμύρια σε εταιρείε που δεν έχουν καμία σχέση με την εκπαίδευση ή την έρευνα και δεν έχουν κανένα λόγο να πάρουν αυτά τα κονδύλια. Ο Υπουργό Γεωργία, ο οποίο ε, γνωρίζει 300 υποθέσει μικρών γεωργών που δεν μπόρεσαν να λάβουν καμία επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί κάποιε μεγάλε εταιρείε ε, παίρνουν τι επιδοτήσει, ενώ θα να τι παίρνουν οι μικροί γεωργοί, Αυτές οι επιδοτήσεις ε, σταμάτησαν και τώρα οι γεωργοί περιμένουν εδώ και χρόνια να λυθεί το πρόβλημά τους δικαστικά. Κάποιοι από τους γεωργούς έχουν ε, πέσει και θύματα ε, βίας. Ο γεωργός Βλάντο Ριμπάρ ε, απειλήθηκε και βρέθηκε νεκρός τέλη του έτους, πέρυσι. Και υπάρχει έρευνα για το φόνο του. Ε, σε, μια τηλεοπτική, σε ένα τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ οι γεωργοί ισχυρήθηκαν ότι τους προσέφεραν επιδοτήσεις, αλλά έπρεπε να πληρώσουν όμως για να πάρουν αυτά τα λεφτά. Έπρεπε να πληρώσουν δηλαδή ε, φακελάκι. Και οι τιμές ήταν γενικά ε, 30.000, για, όταν τους δίνανε 100.000 επιδοτήσεις ή 15.000 ε, δίναν φακελάκι από τις 50.000 που τους δίνανε σε επιδοτήσεις. Λοιπόν, έκανα εγώ μια μικρή έρευνα. 33% του κόσμου έχουν ε, λιγότερη εμπιστοσύνη και πολύ περισσότεροι δεν έχουν καθόλου εμπιστοσύνη. Ρώτησα τον κόσμο πώς αισθάνεται για το γεγονός ότι η έρευνα για τη δολοφονία πήγε στο, στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών. Το 88% αισθάνονται φόβο γι' αυτό. Ε, τους ρώτησαν, ε, θεωρούν ότι ε, υπάρχει διαφθορά στη Σλοβακία. Το 97% είπαν ότι δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη και πιστεύουν ότι υπάρχει διαφθορά. Τον Ιανουάριο του 2019, ο νέος επικεφαλής αστυνομίας είπε ότι η δολοφονία ε, έχει διερευνηθεί κατά το 25% ένα χρόνο μετά τη δολοφονία των ανθρώπων αυτών, του Γιάννη και της Μαρτίνα. Υπάρχει ένα, μια πρόταση για ψήφισμα ε, που έγινε χθες δεχτή. Είναι καλή αρχή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισκέφθηκε τη Σλοβακία, μας έδωσε ελπίδα και έκανε μεγάλη εντύπωση η επίσκεψη αυτή. Αλλά η δουλειά δεν μπορεί να σταματήσει εκεί. Υπάρχει ένα συνέστημα κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλο και μεγαλύτερο στη Σλοβακία. Λόγω αυτού του ανθρώπου, το οποίο, ο οποίος τώρα κατεβαίνει για πρόεδρος. Μην ξεχνάτε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αδιαφορούν, που δεν πιστεύουν ε, που δεν έχουν εμπιστοσύνη στην Ευρώπη και στις αξίες της. Ε, οι επιπτώσεις της διαφθοράς σε εθνικό επίπεδο ε, αλλοιώνουν την άποψη των ανθρώπων και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να δει και να έρθει σε επαφή με τους ανθρώπους, με τους ακτιβιστές και να μην βασίζεται μόνο σε υπαλλήλου και αξιωματούχους στις χώρες. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έρθει πιο κοντά στους ανθρώπους ε, να αισθανθούν όλοι οι άνθρωποι και αυτοί που βρίσκονται χαμηλά στην κοινωνική κλίμακα ότι η φωνή τους μετράει, ότι είναι τμήμα αυτής της κοινωνίας, της δημοκρατίας και ότι έχουν εξουσία και μπορούν για να μπορούν να ελπίζουν στο χώρο αυτό ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφάλειας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ακούτε την ε, απόλυτη αυτή σιωπή στην αίθουσα. Νομίζω ότι μιλάει από μόνη τη. Ε, ήταν ένα σοκ για όλου αυτό το οποίο είπατε. Η κυρία Φρόνσκα τώρα έχει το λόγο εξ ονόματο τη Ευρωπόλ. Καλησπέρα σα. Σα ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και για τη δυνατότητα που δίνετε στην Ευρωπόλ να πάρει το λόγο στη δική σα την Επιτροπή. Η Ευρωπόλ όντω πλάκη στις ε, έρευνες ε, της ε, υπόθεσης αυτής βάσει αιτήματο που απίφθινε η οικία χώρα. Θα ήθελα εδώ πέρα να τονίσω ότι η Ευρωπόλ μπορεί να αναλάβει δράση για να υποστηρίξει ένα κράτος μέλος στο πλαίσιο της έρευνας μετά από αίτημα του συγκεκριμένου κράτους. Υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι η εγκληματική αυτή πράξη αφορά δύο ή περισσότερα κράτη-μέλη. Συνέβη όντω κάτι τέτοιο και όντω έχουμε θεσπίσει μια πολύ θετική συνεργασία και όπως γνωρίζετε η έρευνα για τη δολοφονία αυτή βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Η Ευρωπόλ προφανώς συνεργάζεται με τις Σλοβακικές Αρχές οι οποίες δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο της μικτής ομάδας έρευνας. Δίνουμε τεχνική υποστήριξη προς, τους, προς αρχές της Σλοβεκίας. Η διαδικασία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Τώρα η ερευνητική ομάδα η οποία διερευνά την δολοφονία αυτή έχει πολύ καλές σχέσεις με τους εμπειρογνώμονες της Ευρωπόλ και υπάρχει ένα γενικότερο πνεύμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Είχαμε ανταλλαγή πολλών σημαντικών πληροφοριών, κάναμε ελέγχου και από τις δύο πλευρές και προσπαθήσαμε από επαγγελματικής πλευράς να προωθήσουμε περισσότερο συνεργασία αυτή και οι πυρογνώμονες Ευρωπόλ θεωρούν ότι είναι ιδιαίτερα επιτυχής μέχρι στιγμή αυτή η συνεργασία. Βέβαια, Βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη η όλη έρευνα και βάσει των πληροφοριών που διαθέτω η επέκταση της διάρκειας της κοινής αυτής ερευνητικής ομάδας θα συζητηθεί σύντομα και θα ληφθεί σύντομα μια απόφαση από τις δύο μπλεκόμενες χώρες, τη Σλοβακία και την Ιταλία. Αυτή είναι, αν θέλετε, η οπτική γωνία της Ευρωπόλ μέχρι στιγμής και προφανώς Είμαστε στη διάθεση των ερευνητών για να υποστηρίξουμε σε όλα τα επίπεδα το έργο τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Η κυρία Ούρσκα Μπάβοβιτς μπορεί να πάρει τώρα το λόγο από τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω την αναφέρουσα, την κυρία Παπούντοβα, για την παρουσίαση που μας έκανε, ιδιαίτερα διαφωτιστική μας δώσετε μια σαφέστατη κατάσταση, σαφέστατη εικόνα της κατάστασης που αντιμετωπίσετε στη χώρα σας. Καταρχάς θα ήθελα να κάνω κάποιες γενικές παρατηρήσεις, λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γενικότερα το λεγόμενο ευρωπαϊκό επίπεδο δίνει ιδιαίτερη σημασία στη δικαστική συνεργασία σε εγκληματικές υποθέσεις. Ο λόγο για τον οποίο θεωρήθηκε μάλιστα η κοινωνική βάση για την Ευρωπόλ ήταν ακριβώ αυτό, να καταφέρουμε να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα τη Ευρωπόλ κάθε φορά που θέλει να συντονίσει, να υποστηρίξει και να βοηθήσει καλύτερα τι εθνικέ αρχέ που διερευνούν συγκεκριμένε υποθέσει. Όπω είπατε πολύ σωστά στο πλαίσιο τη παρουσίασή σα, η Βέρα Γιούροβα, η επίτροπό μα, όταν πήγε στη Σλοβακία, τοποθετήθηκε και μίλησε υπέρ της υποστήριξη Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κάλεσε μάλιστα τις σλοβακικέ Αρχές να προχωρήσουν στα παρέτα βήματα προκειμένου να βρεθούν οι πέτοι της δολοφονίας του Γιάνν Κουτσιάκα και της Μαρίνα Κουσνίροβα. Και σας ευχαριστώ πολύ που αναφερθήκατε και στο έργο της Επιτρόπου. Όσον αφορά τώρα την επιχειρησιακή πλευρά, η εκπρόσωπος Ευρωπόλ Μόλις τώρα τόνισε πολλές πτυχές της ε, λειτουργικής αυτής πλευράς. Να δώσω και εγώ κάποια περαιτέρω στοιχεία. Ουσιαστικά η DigiJust, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήρθε σε επαφή με τη Eurojust ζητώντα τη να ενημερωθεί για το πώ έχουν τα πράγματα όσον αφορά τη διερεύνηση τη συγκεκριμένη υπόθεση. Λάβαμε από τη Eurojust κάποιε πληροφορίε ότι όντω βρίσκεται σε εξέλιξη η όλη έρευνα, άρα δεν μπορούν να μα δώσουν συγκεκριμένα στοιχεία για τα πραγματικά περιστατικά. Ωστόσο, η Eurojust επιβεβαίωσε ότι όντω θεσπίστηκε μια κοινή ομάδα ερευνών για τη διερεύνηση των δολοφονιών αυτών και αυτό έχει ανακοινωθεί και από την ίδια τη Eurojust επισήμω, η οποία λέει ότι υποστηρίζει από οργανωτική και τεχνική πλευρά την όλη έρευνα. Τώρα, όσον αφορά το δελτίο τύπου τη ε, Eurojust, η οποία είπε στο πλαίσιο του δελτίου αυτού τύπου ότι και η ίδια Eurojust αλλά και τα εμπλεκόμενα κράτη-μέλη επιθυμούν να συνεχίσουν τη διερεύνηση αυτή. Προφανώς όμως είναι οι αρμόδιες εθνικές αρχές που είναι οι πλέον ε, αρμόδιες για τη διερεύνηση της ε, υπόθεσης αυτής και η Eurojust ουσιαστικά είχε έναν ρόλο συνοδευτικό, υποστηρικτικό. Αυτό είχα να σας πω από τη δική μου την πλευρά. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Οι ευρωβουλευτές τώρα μπορούν να πάρουν το λόγο. Κυρία Μιράντα πρώτη. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να χαιρετήσω την αναφέρουσα και λυπούμεθα για αυτή τη δολοφονία βαθύτατα Εμείς ετοιμάζουμε πληροφορίες για τη σχέση της, μα... μαφίας με την ε, σλοβακική κυβέρνηση και την ε, κακή χρήση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Και για να στείλουμε από εδώ, από την ομάδα μας, ε, στοιχεία για να ευαισθητοποιήσουμε όλο τον κόσμο και να καταδικάσουμε ένα επεισόδιο όπου οι πληροφοριοδότες, οι καταγγέλλοντες κινδυνεύουν πια, μπαίνουν σε δύσκολη θέση. Είναι εκτεθειμένοι και μπορεί να δολοφονηθούν τελικά. Υπ' αυτή την έννοια η Σλοβακία είναι πολύ ψηλά σε ό,τι αφορά την διαφθορά. Ε, είναι από τις τελευταίες χώρες ό,τι αφορά την εμπιστοσύνη του πολίτη προς τις αρχές, υπάρχει κακό κλίμα, ε, κακή διαχείριση από πλευράς κυβέρνησης της κατάστασης ε, αυτής της δολοφονίας. Αυτό είναι φρικτό. Έχουμε αυτό το ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Κομισιόν ετοιμάζει νομοθετικά κείμενα για να προστατεύει τους πληροφοριοδότες, τους whistleblowers. Ε, είναι κρίμα που δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες για αυτή την υπόθεση δολοφονίας. Νομίζω ότι η θέση της Europol ε, είναι σωστή, ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια σε αυτή την ε, περίπτωση, περισσότερες προφορίες. Η ομάδα μας λοιπόν ζητάει να παραμείνει ανοιχτή αυτή η έκθεση, να πάει στη ΛΥΜΠΕ, στην Επιτροπή ε, Πολιτικών Ελευθεριών. Εγώ είμαι σε αυτή την Επιτροπή και η Σοφή, ούτως ώστε να την παρακολουθήσουμε, να δούμε τι συνέχεια θα δοθεί. Γιατί αυτά τα δύο άτομα πλήρωσαν με τη ζωή τους το γεγονός ότι πολεμούσαν ε, κατά της διαφθοράς και υπέρ της αλήθειας. Ευχαριστώ. Yes, thank you. Ευχαριστούμε Σοφίν Βέλτ, έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Παπκούνοβα. Ελπίζω να προφέρω σωστά το όνομά σας. Σας ευχαριστώ για την αφορά σας και για την παρουσίαση που κάνατε. Και όπως είπατε ήδη χθε εγκρίναμε ένα ψήφισμα για τη Σλοβακία και για τη Μάλτα. Και από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια ισχυρή υποστήριξη από όλες τις βασικές, αν θέλετε, πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έτσι ώστε να συνεχίσει η εργασία και μετά την έγκριση του ψηφίσματος αυτού και στην επόμενη κοινοβουλευτική θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γιατί προφανώς το ζήτημα αυτό απαιτεί κάτι πολύ παραπάνω από την έγκριση ενός απλού ψηφίσματος. Είναι, θα έλεγα, μια μακροπρόθεσμη επένδυση την οποία πρέπει να κάνουμε. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν ακόμα ένα-δύο ερωτήματα που θέλω να θέσω προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπόλ. Καταρχάς, η Ευρωπόλ μας είπε ότι ε, εμπλέκεται πλήρω στην όλη διερεύνηση των δολοφονιών. Αν δεν κάνω λάθο, η κοινή ομάδα ερευνών όμω είναι μεταξύ τη Σλοβακία και τη Ιταλία, έτσι δεν είναι. Και η Ευρωπόλ παρέχει τεχνική υποστήριξη. Ωστόσο, επί τη αρχή όμω είχατε και εσεί πρόσβαση στην πλήρη έρευνα, στην πλήρη δικογραφία, έτσι δεν είναι. ότι αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε ακριβώ τι συνέβη με το τηλέφωνο της Κυρία Χόλτσοβα. Πάντω, τώρα που έχει μοιραστεί, αν θέλετε, η όλη έρευνα, ένα τμήμα τη έχει να κάνει περισσότερο με κάποιες αποκαλύψεις ή έρευνες αυτό το τμήμα ουσιαστικά έχει να κάνει πλέον με το Υπουργείο Εσωτερικών, αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών. Στην περίπτωση αυτή η Ευρωπόλ εμπλέκεται τελικά μόνο στη διερεύνηση της δολοφονίας, ενώ όλες οι υπόλοιπε ε, έρευνε σα διαφεύγουν. Αυτή τη στιγμή δεν έχετε καμία πρόσβαση εσεί στι υπόλοιπε παράλληλε έρευνε που λαμβάνουν χώρα. Αυτό θα ήθελα να μου πει η Ευρωπόλ. Τώρα απευθύνομαι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατά την άποψή μου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να ηγείται περισσότερο τη όλη διαδικασίες. Αναφερθήκατε σε κάποιες απάτες που έχουν γίνει με τα γεωρικά ταμεία. Τέτοια φαινόμενα έχουμε δει και σε άλλες χώρες. Μαζικές απάτες όμως. Αναφερόμαστε σε δισεκατομμύρια ευρώ. Και αυτό μας το καταγγέλουν και πολλοί γεωργοί με τους οποίους ήρθαμε σε επαφή στην Πρατισλάβα. Μας λένε ότι οι έλεγχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι καθαρά γραφειοκρατικοί και επιφανειακοί. Ουσιαστικά δεν πάνε επί τόπου και δεν συνομιλούν επί τόπου με τους ηθήνοντες και δεν επαληθεύουν τελικά αν τα στοιχεία που τους δίνουν οι Σλοβαϊκές Αρχές είναι όντω έγκυρα ή αν τελικά σας κορυδεύουν οι Σλοβαϊκές Αρχές. Αυτό δεν το επαληθεύεται. Ξέρω ότι η κυρία Γκρέσλε από την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού ασχολείται πάρα πολύ με το ζήτημα αυτό και νομίζω ότι η κυρία Γκρέσλε δεν είναι πρώτο σε καμία περίπτωση να αφήσει την κατάσταση αυτή να της διαφύγει και είμαι σίγουρη ότι θα κάνει κάθε τι το δυνατό προκειμένου να συνεργαστεί όχι μόνο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά ακόμα και με την Όλαφ, ακόμα και με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία του να αυτή συσταθεί. Τέλος, πολλά θα μπορούσε να πει κανεί για τη Σλοβακία. Ένα πράγμα πάντω, το οποίο με έναν πογοτεύει όλο ιδιαιτέρω, είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει όλη αυτή η μεταπίδηση από τη μία θέση στην άλλη. Παρετείται ο κύριο Φίκο και ξαφνικά εμφανίζεται πάλι σε μία άλλη θέση. Το ίδιο έκανε και ο κύριο Γκασπάρ και πολλοί άλλοι πολιτικοί θύνοντε. Και γνωρίζουμε ότι μολονότι μεταπηδούν από τη μία θέση στην άλλη, εξακολουθούν και κινούν τα ενία. Ο κύριο Πελεγκρίνη, νέο πρωθυπουργό, θα είναι στην επόμενη ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο και ελπίζω ότι κάποιο μα ακούει εδώ από τι Ευρωπαϊκέ Αρχέ και α του διαβιβάσει το μήνυμα. Περιμένουμε από τον κύριο Πελεγκρίνη την επόμενη, τον επόμενο μήνα να στείλει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Τι είναι πιο σημαντικό η φιλία του με τον κύριο Φίκο και η συμμετοχή στο πολιτικό του κόμμα ή περισσότερο η ευρωπαϊκή, αν θέλετε, διάσταση και η πολιτική του ομάδα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αν πραγματικά ενδιαφέρεται τελικά για την προάσπιση των συμφερόντων των πολιτών του. Σε αυτό το βασικό ερώτημα θα κληθεί να απαντήσει όταν έρθει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Δύο λεπτά τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δύο λεπτά στην Ευρωπόλ προκειμένου να ολοκληρωθεί η συζήτηση. Ας ακούσουμε όμως πρώτα την κυρία Εύη, μετά την κυρία Εστέρα Φαραγκούτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Παίρνω και εγώ το λόγο για αυτή την αναφορά. Θέλω να δείξω αλληλεγγύη στις οικογένειες του Γιάννη και της Μαρτίνα για αυτά που ζου, ζουν τώρα και για αυτά που ζήσανε. Ευχαριστώ την αναφέρουσα που μας παρουσίασε σήμερα αυτή την αναφορά και αυτή την συγκλονιστική περιγραφή του τι συνέβη. Θέλω να δώσω σημασία να σταθώ σε ένα στοιχείο της υπόθεσης αυτής. Γιατί οι έρευνες που έγιναν έδειξαν ότι υπάρχουν στενότατες σχέσεις ανάμεσα ε, στους παράγοντες του Σπίκου και στην Ντράγκετα. Η Ντράγκετα δραστηριοποιείται στην ε, Σλοβακία και έχει και στενούς δεσμούς και όλο αυτό ανεβαίνει ως κατευθείαν το Φίκο. Ο εισαγγελέα της, της Καλάμπρια, λίγες μέρες μετά τη θολοφονία του Γιάννη και της Μαρτίνα, όταν ξεκαθαρίστηκαν περισσότερο η συμμετοχή της Ντράγκετα και με, τις, με τους ανώτατους ηθήνοντες και πολιτικούς της Σλοβακίας είπε ότι πολύ εύκολα έκανε παιχνίδι η Ντράγκετα στην Σλοβακία και πολύ εύκολα διείσδησε γιατί ακριβώς υπήρχε απουσία, υπήρχε ε, ανισότητα και δεν υπήρχαν και εργαλεία για να καταπολεμηθεί η μαφία στο Σλοβακικό κράτος. Όπως σε πολλά άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Υπάρχει ε, το αδίκημα το, για δημιουργία συμμορίας ε, με σκοπό τη διάπραξη μαφιόζικων ε, εγκλημάτων. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να έχουμε πιο προηγμένους κανόνες για να καταπολεμήσουμε το οργανωμένο έγκλημα μαφιόζικης απόχρωσης. Είναι απαραίτητο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναγνωρίσουμε αυτό το αδίκημα, ότι δηλαδή συμπίζει κανείς συμμορία με σκοπό να διαπράξει μαφιόζικα εγκλήματα. Ε, αυτά ε, είναι εγκλήματα που υπάρχουν στην Ήπειρό μα ε, με διεθνεί τάσει. Στηρίζω λοιπόν απόλυτα αυτή την αναφορά. Συμφωνώ με τα ερωτήματα που έγιναν από τη συνάδελφο και εγώ περιμένω να ακούσω μια απάντηση. Νομίζω όμως ότι αυτή, αναφο... ότι αυτή η Επιτροπή Αναφορών μπορεί να κάνει περισσότερα πράγματα. Δεν ξέρω αν θα έχουμε το χρόνο. Αλλά ακόμα και τελευταία στιγμή. Έτσι θα μπορούσαμε κάπου να χωρέσουμε μία ερευνητική επιτροπή, ας πούμε, ή διερευνητική καλύτερα επιτροπή, της Επιτροπής ΠΕΤΗ. Αισθάνομαι πάρα πολύ κοντά σε όλους τους α, Σλοβάκους, τους τίμους Σλοβάκους πολίτες ε, που δίνουν μάχη. Η Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ρενάτα Παπκούνοβα, την α, αναφέρουσα ελπίζω να μην σκότωσα το όνομά σας, και την ε, Επιτροπή και την Κατερίνα Φλέκοβα, ε, που εκπροσωπεί τη Europol, το, θεσμικό, το τμήμα θεσμικών υποθέσεων της Europol. Τα τελευταία χρόνια είχαμε μια διαδοχή ε, δολοφονιών δημοσιογράφων, ερευνητών δημοσιογράφων, που έγιναν στη Μαλτία, στη Σλοβακία, στη Βουλγαρία, στη Σουηδία η ήπειρο των Αξιών και της Ειρήνης, που είναι το παράδειγμα δημοκρατίας και του κράτους δικαίου και της ευημερίας, ξαφνικά ε, στυλιτεύεται με αυτόν τον τρόπο. Ε, η ερώτηση είναι, κάνουμε ό,τι μπορούμε, μήπως μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Επομένως, ε, γι' αυτό είναι πολύ κέρια η αναφορά. Έγιναν συζητήσει ε, στο Κοινοβούλιο για αυτό το θέμα και στο Στρασβούργο ήρθε η οικογένεια του Καρουάνα, για, της ε, Γκαρουάνα μάλλον για την ε, υπόθεση της Μάλτας. Ε, συζητήθηκε και στην υπόθεση ε, πολιτικών ελευθεριών. Το βασικό είναι να συνεργαστούμε πολύ στενά με τις σλοβασικές αρχές ε, για να υπάρχει εγγύηση ε, ουδετερότητας και αμεροληψίας. Υπάρχει συνεργασία για ποινικά θέματα, ε, είναι πολύ σημαντική αυτή. Ξέρω ότι δεν έχουμε πληροφορίες, γιατί υποτίθεται είναι στις τελικές φάσεις η έρευνα, αλλά έχουμε μια εγγύηση γιατί η Europol εμπλέκεται. Το βασικό όμως είναι να μείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε ούτως ώστε να βοηθήσουμε ό,τι μπορούμε και για να βοηθήσουμε τις αρχές της Europol, να βοηθήσουμε την Κομισιόν, ό,τι μπορείτε να σκεφτείτε. Γιατί εμείς είμαστε μια επιτροπή που προσπαθεί να βοηθήσει. Προσπαθούμε να ασκήσουμε πίεση και να αφυπνίσουμε συνειδήσεις. Ας κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ούτω να μην μείνει κανένας άεργο και δεν κάνει κάτι που θα μπορούσε να κάνει. Όχι μόνο για τη Σλοβακία και τις ε, οικογένειες των θυμάτων που τη στηρίζουμε, αλλά για όλη την Ευρώπη και για αυτό που εκπροσωπεί η Ευρώπη. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Δεμέρα τώρα το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κάποιες σκέψεις. Καταρχάς, πολύ θετική αξιολόγηση της έκθεσης αυτής της Ρενάτα και του θάρρους της που ήρθε εδώ και την παρουσίασε σε μια ανοιχτή επιτροπή. Που την ακούνε όλοι. Δεύτερον, έχω μια αμφιβολία. Μια υποψία ορθολογικού χαρακτήρα. Η υποψία και η αμφιβολία είναι ότι η κυβέρνηση των κυβερνήσεων οι κυβερνήσει της Σλοβακία χρησιμοποίησαν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα που είναι τόσο αξιόπιστα όπως η Eurojust, η Europol, για να αποκτήσουν άλοθη, ενώ στην πραγματικότητα ε, δεν θέλουν μια διαφανή ε, δικαστική έρευνα, αλλά για να αποκτήσουν άλοθη ότι πραγματικά ε, διεξάγεται μια τέτοια διαφανής έρευνα. Θα έπρεπε η Eurojust και η Europol να τους δώσει, να τις υποχρεώσει να δώσουν πιο ακριβείς πληροφορίες. Γιατί όλοι ξέρουν ότι συχνά μιλάμε για τέτοιες περιπτώσεις για επιμελητιακή ή πρακτική στήριξη. Όλοι ξέρουμε τι είναι αυτή η πρακτική στήριξη. Μπορεί να είναι να πληρώσουμε, ας πούμε, βενζίνη για τα αυτοκίνητα, ας πούμε. Έτσι. Και άλλα πράγματα. Αλλά στην περίπτωση της Europol, εγώ έχω μεγάλη εμπιστοσύνη. Την πιστεύω απόλυτα. Αν χρειαστεί να δημιουργηθεί μία μεικτή ομάδα, ε, δηλαδή ε, πρόσωπα, προσωπικό από δύο διαφορετικά κράτη να εμπλακούν σε μία έρευνα και να πάνε στη Σλοβακία, καλό θα ήταν. Άκουσα το σχόλιο της Κατερίνα. Η παρουσίαση αυτή είναι σύντομη και συμβατική. Εγώ θα ήθελα μία πιο λεπτομερή, πιο ακριβή παρουσίαση. για τις ποινικέ ε, έρευνες. Γιατί. Το βασικό είναι βέβαια να πιέσουμε τη Σλοβακία να κάνει αυτή την ε, εγκληματική έρευνα. Ε, η Σλοβακία είναι ο πρωταγωνιστής. Δεν είναι η Κομισιόν, δεν είναι κανένας άλλος. Κάποιο αρμόδιο στη Σλοβακία είπε ότι έχουμε διερευνήσει το 25% τη υπόθεση. Πώ μετράτε αυτό το 25%, με ποιο θερμόμετρο, α πούμε, μετράτε αυτό το νούμερο, α πούμε. Φτάσατε στο 25% τη έρευνα. Τι θέλω να σας πω με όλα αυτά. Θέλω να σας πω ότι έχω αμφιβολίες. Δεν θέλω να χρησιμοποιούν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα που έχουν καταπληκτικό ρέκορντ, φοβερή ε, αξιοπιστία, ως άλοθη για να δείξουν στην κοινή γνώμη ότι πραγματικά υπάρχει διαφάνεια και σοβαρή έρευνα. Φοβάμαι ότι δεν υπάρχει καμία διαφάνεια, δεν υπάρχει δέσμευση των σοβακικών αργών, αρχών να κάνουν σοβαρή έρευνα. Σας ευχαριστώ πολύ. Δύο και δύο λεπτά αντίστοιχα ε, από την Europol, κυρία Μερόσκα. Σας ευχαριστώ πολύ. και ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη συνεχιζόμενη υποστήριξη του προς την Europol. Μία σύντομη απάντηση. Όπως έχω αναφέρει στο παρελθόν, η Europol αντιδράει σε αιτήματα των κρατών μελών. Αναφέρθηκε από τον συνάδελφο από την Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης ότι ε, τέτοιες ε, περιπτώσεις αποτελούν, η ποινική δίωξη αποτελεί θέμα των εθνικών αρχών. Η Europol παρέχει βοήθεια, υποστήριξη στις ε, εθνικές αρχές και είμαστε πάντα διατεθειμένοι να εντείνουμε τις προσπάθειές μας καθότι αυτή η υπόθεση είναι υπόθεση προτεραιότητας για τον οργανισμό μας. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρία Βούπιτς, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο. Από ό,τι καταλαβαίνω, το ερώτημα ήταν του συναδέλφου. Ζητώ συγγνώμη, δεν έχω συγκρατήσει το όνομά σας. Um, it's regarding the corruption in... Ερώτηση της Σοφίας ήταν που είχε να κάνει με διαφθορά όσον αφορά τα γεωργικά ταμεία και ε, γίνονται προσπάθειες για να καταπολεμηθεί η διαφθορά. Ένα από τα μέτρα αυτά είναι ο ορισμός αρμόδιας αρχής που θα ασχολείται με τέτοιες ε, υποθέσεις. Αυτά από μένα. Πολύ σύντομα, κυρία Νετφέλ. Δεν καταλάβα από την απάντησή σας εάν θα συμμετέχετε και στις άλλες έρευνες. Είπατε ότι δεν είναι δική σας αρμοδιότητα ή είναι κάτι που ανήκει σε άλλο Υπουργείο, αλλά αυτό ακούγεται σαν να θέλετε να αποκλείσετε την Ευρώπη από ε, τις έρευνες, ε, σαν να μην θέλουν να δείτε κάποια πράγματα. Επίσης, όσον αφορά τις, ε, ε, τις ε, σλοβακικές αρχές, από ό,τι κατάλαβα, η προθεσμία λήγει στις 18 Απριλίου. Θα παραταθεί, έχει ζητηθεί η παράταση. Επιτρέψτε μου να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Ζητήθηκε από τη Europol να παράσχει υποστήριξη στις έρευνες της δολοφονίας. Ο οργανισμός μας παρέχει συνεχώς την σχετική υποστήριξη όσον αφορά την ε, παράταση για την ε, κοινή ε, διερευνητική ομάδα, την JIT. Αυτό είναι θέμα που αφορά την Σλοβακία και την Ιταλία και τις άλλες χώρες που συμμετέχουν. Η σχετική απόφαση θα ληφθεί μέσα σε επόμενες εβδομάδες. Δεν έχουμε ακόμη σχετικές πληροφορίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου να συνοψίσω μια πιθανή απόφαση από τη δική μας πλευρά. Θα παραμείνει ανοιχτή η αναφορά. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Δεύτερον, θα στείλουμε επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα της ζητήσουμε να παρακολουθήσει την διενέργεια των ερευνών στην Σλοβακία. Τρίτον, θα στείλουμε επιστολή στην κυβέρνηση της Σλοβακίας. λέγοντας ε, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να παρακολουθεί τη διενέργεια ε, των ερευνών ε, για τη δολοφονία αυτή. Επίσης θα ενημερώσουμε τους συναδέρφους μας στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ για την αναφορά αυτή και θα τους συζητήσουμε να συντονίσουμε τις ενέργειές μας στον τομέα αυτών στο μέλλον. Και πέμπτον, και αυτό είναι κάπως ασυνήθιστο, προτείνω η Επιτροπή Αναφορών να αποφασίσει στο δεύτερο μισό του έτους αυτού ε, να πραγματοποιήσει η δεύτερη αποστολή στην Σλοβακία. Αυτό φυσικά θα γίνει μετά τις ευρωεκλογές, αλλά πιστεύω ότι και η μελλοντική Επιτροπή Αναφορών θα πρέπει να ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Φαίνεται να υπάρχουν πολλά εκρεμή ζητήματα τα οποία δεν μπορούμε να απαντήσουμε αυτή τη στιγμή. Ελπίζω να διαλευκανθεί με επαγγελματικό τρόπο αυτή η δολοφονία. Νομίζω όμως ότι και οι μελλοντικοί μας συνάδελφοι θα πρέπει να ασχοληθούν με το θέμα. Συμφωνείτε με την πρότασή μας. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ. Η επόμενη αναφορά έχει αριθμό 490 του 2018 από τη Ρουμανία. Με ενημερώνουν ότι δεν είναι παρόν ο αναφέρον. Θα παρακαλούσα τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης ε, να μας ε, εξηγήσει τη θέση της. Παρακαλώ. Ε, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Καταρχάς, να σας ζητήσω εκ των προτέρων συγγνώμη, γιατί από όσο κατάλαβα η απάντηση ακόμα δεν έχει φτάσει στην Επιτροπή Αναφορών, γιατί ακόμα μεταφράζεται βασικά. Επομένως, θα ήθελα να σας διαβάσω εδώ πέρα την προτινόμενη απάντηση, η οποία θα σας διαβαστεί και επισήμως, ελπίζω σύντομα. Όπως ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 23 Απριλίου μια πρόταση για μια οδηγία για την προστασία των ε, καταγγελόντων ε, της παραβίασης ε, του νοσιακού δικαίου. Αυτή τη στιγμή ε, περάσει στο εθνικό δίκαιο η πρόταση αυτή θα διασφαλίσει ένα πολύ ψηλό επίπεδο προστασία για του κατακέλλοντε, ε, οι οποίοι αναφέρουν παραβιάσει ε, του νοσιακού δικαίου σε συγκεκριμένου τομεί πολιτική και θα υπάρχει νέο επίπεδο προτύπων προστασία. Ανάμεσα στα πρότυπα αυτά, στην πρόταση προβλέπεται ότι οι εργοδότε του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα θα φέρουν συγκεκριμένους, ε, συγκεκριμένες ευθύνες και θα έχουν συγκεκριμένους διάβλους προκειμένου να υποβάλουν πληροφορίες στον ιδιωτικό ή τον ε, δημόσιο τομέα προς τις ε, αρμόδιες αρχές. Αν δεν υπάρχουν τώρα οι διάβλοι αυτοί, τότε θα μπορούν άμεσα να απευθύνονται στις αρχές αυτές οι ίδιοι κατακέλλοντες και θα πρέπει να δείτε συνέχεια, συνέχεια στην καταγγελία αυτή. Έπειτα, θα πρέπει να ενημερώνεται και ο ίδιος ο καταγγέλων και να του εξηγείται ακριβώς ποια δράση αναλαμβάνεται από την αρμόδια εθνική αρχή. Μια άλλη τώρα σημαντική υποχρέωση που απορρέει από την πρόταση οδηγίας είναι η διατήρηση της εμπιστευτικότητας σε όλα τα στάδια της υποβολής πληροφοριών. Στην πρόταση οδηγίας προβλέπεται μία σαφής διάταξη κατά τον αντι και θα προβλέπεται συγκεκριμένο κατάλογο μέτρων υπεράσπιση των ε, καταγγελόντων. Μέσω των ελάχιστων αυτών προτύπων θα ενισχύεται η εφαρμογή του νησιακού δικαίου και θα ενισχύεται η λογοδοσία, η διαφάνεια και η ελευθερία τη έκφραση. Καθότι ένα από τα μέτρα είναι η προστασία των ε, ένα από τα μέτρα προστασία αφορά του καταγγέλου τη εκείνη, οι οποίοι στρέφονται κατά των ίδιων των δημοσίων αρχών. Είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι για την λειτουργία των δημοκρατικών κοινωνιών είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνονται καταγγελίε αυτέ και γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται και με το Κοινοβούλιο σα αλλά και με το Συμβούλιο προκειμένου να εγκριθεί μία πρόταση ή δυνατόν πριν το τέλος της τρέχουσας θητείας. Καθώ όμω η πρόταση αυτή οδηγία δεν έχει ακόμα εγκριθεί, αυτό το οποίο έχουμε είναι η τομεακή νομοθεσία που προβλέπει προστασία των καταγγελόντων και κυρίω έχει να κάνει με τι χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε και την καταπολέμηση νομοποίηση ε, εσόδων παράνομε δραστηριότητε. Δυστυχώ αυτή τη στιγμή δεν μα σε θέση εμεί να πούμε αν η συγκεκριμένη αφορά εμπίπτει στην τομεακή αυτή νομοθεσία που υφίσταται αυτή τη στιγμή. Και αυτή τη στιγμή ε, ισχύει μόνο αυτή η τομεακή νομοθεσία. Δεν μπορούμε να πούμε αν εφαρμόζει την νομοθεσία αυτή τελικά η Ρουμανία και ενέχεται στην όλη επίθεση κατά αυτόν τον τρόπο και ο Ευρωπαϊκό Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που όμω δεν μπορεί να εφαρμοστεί συγκεκριμένη περίπτωση. Σε τέτοιε λοιπόν περιπτώσει όπου δεν υπάρχει το απαραίτητο νομικό πλαίσιο για την προστασία των καταγγελόντων, να στα κράτη-μέλη να προβλέπουν ότι προστατεύονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και οι αναφέροντες, ε, οι καταγγέλλοντες μπορούν να προσφεύγουν στα εθνικά δικαστήρια, αλλά και στον εθνικό συνήγορο του πολίτη, καθότι ο αναφέρον εδώ πέρα αναφέρεται και σε κακοδιαχείριση εκ μέρους της ε, κυβέρνησης. Τώρα, όσον αφορά το εργατικό δίκαιο, να δώσω το λόγο στη συνάδελφό μου από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε αφορά την ασφάλεια στη δουλειά, αναφέρεται αυτό τον αναφέροντα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα εκτεταμένο νομοθετικό σώμα για προστασία στους εργαζόμενους εναντίον όλων των κινδύνων που αντιμετωπίζουν στο χώρο εργασίας τους. Η ιδιαίτερη σημασία είναι η, το βασικό νομοθετικό εργαλείο που έχουμε, την οδηγία δηλαδή 18 931 που είναι μια οδηγία πλαίσιο και που παρουσιάζει τις ε, γενικέ αρχέ προστασία και την υποχρέωση του εργοδότη να εξασφαλίσει την ασφάλεια και την υγεία του εργαζόμενου από κάθε άποψη και από σε όλους τους τομείς, ιδιωτικό δημόσιο, σε όλους τους τομείς δραστηριότητα και καλύπτει όλους τους κινδύνους ε, κοινωνικούς, ψυχολογικούς, παρενόχληση, harassment. Δηλαδή υπάρχει και μια ειδική διάταξη στην οδηγία, το άρθρο 11.4 που προβλέπει ότι οι εργαζόμενοι, οι εκπρόσωποι, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων ε, δεν θα πρέπει να έρχονται σε, να είναι σε επιζήμια θέση, σε μειονεκτική θέση, λόγω της ε, συμμετοχής τους σε μέτρα που μπορούν να επηρεάσουν ουσιαστικά την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Από την αναφορά Δεν υπάρχει ισχυρισμό ότι στη ρουμανική νομοθεσία θα υπάρχει πρόβλημα και δεν θα ευθυγραμμιστεί αυτή με την ε, ενωσιακή νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασία. Οι ενωσιακέ οδηγίε, όπω ξέρετε, πρέπει να ενσωματώνται στην εθνική νομοθεσία και απόκειται σε εθνικέ αρχέ από εκεί πέρα να εφαρμόσουν ε, και να παρακολουθήσουν την εφαρμογή των εθνικών διατάξεων που εφαρμόσουν εθνική νομοθεσία αυτές τις ε, ευρωπαϊκές οδηγίες και αν υπάρχουν προβλήματα ε, γίνονται, υπάρχουν εθνικές διαδικασίες προσφυγής και ρυθμίζονται από τις εθνικές αρχές. Η Κομισιόν για θέματα υγείας και ασφάλειας πιστεύει, ε, πιστεύουν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι το θέμα αυτό πρέπει να ρυθμιστεί από τις εθνικές αρχές. Η σύστασή μου, γιατί δεν βλέπω άλλους συναδέλφους, είναι η εξή. Να στείλουμε μια ενημέρωση στον αναφέροντα με βάση την παρουσίαση που κάνατε σήμερα και εν συνεχεία να κλείσουμε την αναφορά αυτή. Γιατί δεν υπάρχουν νέα στοιχεία. Συμφωνείτε? Πολύ ωραία, ευχαριστώ. Και τώρα έχουμε την τελευταία αναφορά για την πρωινή συνεδρίασή μας, που είναι η αναφορά 580 του 2018 Τώρα, θέλετε να μιλήσετε μισό λεπτό, μισό λεπτό. Είναι μία αναφορά από τον κύριο Αθανάσιο Κικινή, Έλληνα. Έχετε το λόγο, Καλώ ήρθατε καθώς, και έχετε το λόγο για πέντε λεπτά. Καλημέρα σε όλους και ευχαριστούμε πολύ που δεχτήκατε να είμαστε εδώ παρόντες και να εκφράσουμε την αναφορά μας. Είμαι ο Θανάσης Χικινής, πρόεδρος Δασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος και είμαστε εδώ μαζί με το Προεδρείο της Δασκαλικής Ομοσπονδίας. Ε, εκπροσωπούμε τους 80 περίπου χιλιάδες εκπαιδευτικούς που εργάζονται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στα νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία και ειδικά σχολεία της Ελλάδας και η αναφορά που καταθέτουμε έχει να κάνει με το καθεστώς εργασίας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Πρόκειται για εκπαιδευτικούς οι οποίοι είναι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου που κάθε χρόνο προσλαμβάνονται από το Σεπτέμβριο την έναξη δηλαδή της σχολικής χρονιάς και κατά τη διάρκεια της και απολύονται στις 21 Ιουνίου. Είναι εργαζόμενοι οι οποίοι εξαιτία των πολλών χρόνων που δεν έχει γίνει ούτε ένας διορισμός μόνιμου εκπαιδευτικού στην Ελλάδα για περίπου 10 χρόνια τώρα καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Εργάζονται σε θέσεις που έπρεπε κανονικά να καλύπτονται από μόνιμο προσωπικό εργάζονται σε αυτές τις θέσεις έχοντας την αγωνία κάθε χρόνο εάν θα προσληφθούν, γιατί δεν είναι σίγουρο ότι θα το πετύχουν, έχοντας την αγωνία σε ποιο τόπο θα εργάζονται, γιατί δεν γνωρίζουν ότι δεν εργάζονται στον ίδιο χρόνο, κάτι που κάνει εξαιρετικά κακό και στους ίδιους, αλλά και στο εκπαιδευτικό σύστημα που έχει ανάγκη από σταθερό εκπαιδευτικό προσωπικό, Πολλέ φορέ δεν έχουν τη δυνατότητα καν να κάνουν οικογένειε εξαιτία των πολλαπλών μετακινήσεων και όταν το πετυχαίνουν, πολύ συχνά ζουν μακριά από αυτού χωρισμένοι μεταξύ του στην ουσία, αφού μπορεί να είναι και οι δύο αναπληρωτέ εκπαιδευτικοί ή ο ένα να μετακινείται. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι οι εκπαιδευτικοί αυτοί υφίστανται άνηση μεταχείριση και άδικη μεταχείριση. Πρόκειται για σαφή παραβίαση της κοινοτικής οδηγίας 1990 του 70 αφού Καμία προστασία δεν παρέχεται σε αυτό το προσωπικό, καμιά πρόβληση δεν υπάρχει ικανή για να αποτρέψει καταχρήσει όπω ορίζει η οδηγία, δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί δεν ξέρουν πού και αν θα εργαστούν κάθε χρόνο. Οι αναπληρωτέ και ορομοί εκπαιδευτικοί λαμβάνουν αποδοχέ κατώτερε των μόνιμων συναδέλφων του, αφού αν και παρέχουν την ίδια χρονικά και ποσοτικά εργασία, στην πραγματικότητα λαμβάνουν αποδοχέ μόνο για το διάστημα τη σύμβασή του, σε αντίθεση με του μόνιμου που αμείβονται καθ' τη διάρκεια του έτου. Μένουν με λίγα λόγια για του μήνε στου οποίου δεν δουλεύουν απλήρωτοι και τρίτον, και πάρα πολύ σημαντικό, οι συνάδελφοι αυτοί, αν και παρέχουν τι ίδιε ακριβώ υπηρεσίε με αυτέ που παρέχουν και οι μόνιμοι συνάδελφοί του, έχουν τελείω διαφορετική αντιμετώπιση σε επίπεδο συνθήκων εργασία. Είναι χαρακτηριστικό να το αναφέρουμε ότι ένα μόνιμο εκπαιδευτικό δικαιούται αναρωτική άδεια με αποδοχέ τόσων μηνών όσα είναι και τα έτη τη υπηρεσία του, υπολογιζόμενη και τη αναγνωρισμένη προπηρεσία του, ενώ οι αναπληρωτέ συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικοί δικαιούνται συνολικά 15 ημέρε αναρωτική άδεια με αποδοχέ κατά τη διάρκεια τη σύμβασή του και διατρέχουν, αν ξεπεράσουν αυτό το όριο, να απολυθούν για τη χρονιά την οποία έχουν προσληφθεί. Μπορεί εύκολα να καταλάβει κανεί ότι ένα αναπληρωτή εκπαιδευτικό, ο οποίο χρήζει μεγαλύτερη άδεια λόγω ατυχήματο ή σοβαρή ασθένεια, θα λάβει μόνο 15 μέρε από αυτήν και συνεχεία θα λυθεί η σύμβασή του, ενώ είτε στην καλύτερη περίπτωση θα πάψει να αμείβεται και φυσικά έχουμε διαφορετική αντιμετώπιση σε όλα τα επίπεδα των δικαιωμάτων και σε άδειε μητρότητα, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά και σε, ακόμη και στι διαδικασίε λειτουργία του σχολείου, πολύ πρόσφατα αποκλείστηκαν οι αναπληρωτέ εκπαιδευτικοί από το δικαίωμα να ψηφίσουν στη διαδικασία που υπήρξε για το ποιοι θα είναι διευθυντέ ή υποδιευθυντέ στι σχολικέ μονάδε. Είχαν διαφορετική αντιμετώπιση σε επίπεδο δικαιωμάτων. Ω δασκαλική ομοσπονδία, εκπροσωπώντα αυτού του συναδέλφου και με δεδομένο με βάση την παραβίαση τη κοινοτική οδηγία και την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου το 2014 που αφορούσε ακριβώ την ίδια περίπτωση με του συναδέλφου τη Ιταλία, όπου κρίθηκε σε αυτή την απόφαση του δικαστηρίου ότι είναι αντίθετη στο δίκαιο τη Ένωση η Ιταλική και σαφώ και η Ελληνική στην περίπτωσή μα ρύθμιση για τη σχέση εργασία ορισμένου χρόνου στον κλάδο τη εκπαίδευση, και δεν είναι δικαιολογημένη η απεριόριστη ανανέωση των συμβάσεων αυτών για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών στα δημόσια σχολεία, ζητάμε το αυτονόητο. Το να υπάρξουν μόνιμοι διορισμοί, διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών στην στο σύνολο τη εκπαίδευση, οι άνθρωποι αυτοί να δουλέψουν σε σταθερέ θέσει, να καλυφθούν όλε οι ανάγκε τη εκπαίδευση και φυσικά όσοι συνεχίζουν να εργάζονται ω αναπληρωτέ να έχουν τα ίδια δικαιώματα και όχι υποβαθμισμένη θέση μέσα στο δημόσιο σχολείο. Θα είναι μια απόφαση η οποία θα αποκαταστήσει τη δικαιοσύνη, το αίσθημα δικαίου σε σχέση με αυτού του ανθρώπου και θα συμβάλλει πάρα πολύ στην ε, άνοδο του επίπεδου τη εκπαίδευση στην Ελλάδα, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί έχουμε να κάνουμε με παιδιά που είναι το μέλλον τη χώρα και τη Ευρώπη. Σα ευχαριστώ πολύ. Θα παρακαλούσα την κυρία Σέκιμπαρκ από την Γενική Διεύθυνση Απασχόληση ε, να μας ε, μιλήσει για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και τον αναφέροντα που έθεσε το θέμα. Όπως ακούσαμε, ανησυχεί σχετικά με την οδηγία συγκεκριμένου χρόνου και ιδιαίτερα τη ρήτρα 4 που έχει να κάνει με τη ρήτρα μη διάκρισης ε, των εργαζομένων ε, με σύμβαση ορισμένου χρόνου σε σχέση με τους μονίμους. Επίσης, ε, σχετικά με τη ρήτρα 5 που στόχο έχει να εμποδίσει την κατάχρηση του μέσου των συμβάσεων ορισμένου χρόνου για να καλυφθούν μόνιμες λύσεις. Δεν έχει εφαρμοστεί δηλαδή σωστά η οδηγία όσον αφορά τους ε, δασκάλους ε, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα. Σημειώνουμε αυτά που μας είπε ο αναφέρον όσον αφορά το ε, σημαντικό χρονικό διάστημα που αναφέρεται εδώ πέρα. Κάποιες ε, συμβάσεις ε, ανανεώνονται από το 2002 και επίσης φαίνεται ότι όσον αφορά τις άδειες, τον αριθμό ημερών και την αμοιβή, ότι γίνεται διάκριση σε σχέση με τους μονίμους υπαλλήλους. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να εξετάσει το πώς ε, έχουν εφαρμοστεί οι ρήτρες αυτές στην Ελλάδα όσον αφορά τους δασκάλους στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η κυρία Σοφία Σακοράφα και ο κύριος Ζαριανόπουλος από την Ελλάδα ε, έχουν στείλει επιστολή όπου στηρίζουν την αναφορά αυτή. Ο κύριος Μαριάς, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Βεβαίως η πλήρης υποστήριξη των ετοιμάτων της ΔΟΕ από τους ευρωβουλευτές είναι σημαντική, αλλά κυρίως πρέπει να γίνεται εδώ, στην Επιτροπή. Διαφορετικά και εμείς από την Ελλάδα θα στέλναμε αγωνιστικούς χαιρετισμού και συμπαράσταση στον καθέναν. Αλλά η εργασία και η παρουσία είναι εδώ, παρότι αντιλαμβάνουμε ότι πολλοί αγωνιούν ενδεχόμενα για την επανεκλογή τους στο επόμενο χρονικό διάστημα. Πρόκειται για μια καραμπινάτη περίπτωση παραβίασης της οδηγίας ε, η οποία ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Την οδηγία 1999 του 70. Τι λέει η οδηγία αυτή δύο πράγματα. Πρώτον, όταν υπάρχουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, δεν πρέπει οι εργοδότες, είτε είναι το δημόσιο είτε είναι ο ιδιώτης, να χρησιμοποιεί συμβάσεις ορισμένου χρόνου, προκειμένου να καλύπτει αυτές τις ανάγκες, αλλά ιδίως όταν πρόκειται για το δημόσιο, θα πρέπει να προσδιορίζει τέτοιες λύσεις οι οποίες να μόνιμοποιούν την απασχόληση του προσωπικού. Και δεύτερον, δεν πρέπει οι εργαζόμενοι με ορισμένο χρόνο να έχουν λιγότερα δικαιώματα από αυτούς οι οποίοι απασχολούνται στην ίδια θέση. Εδώ λοιπόν τι έχουμε. Κλασική περίπτωση του ελληνικού δημοσίου όπου στην εκπαίδευση από τους 80.000 εκπαιδευτικούς στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στα νηπιαγωγεία οι 22.000 είναι όμοιροι. Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι κάθε χρόνο αγωνιούν για το αν θα τους ανανεωθεί η σύμβαση, εργάζονται από την έναρξη του σχολικού έτους μέχρι τις 21 Ιουνίου, απολύονται και μετά περιμένουν να δουν αν θα ξαναπροσληφθούν, πιθανόν όχι στην ίδια περιοχή, σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Ενώ υπάρχουν διαπιστωμένες οι και διαρκείς ανάγκες. Και αυτό το κάνουν βεβαίως και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο ελληνικό δημόσιο και σε άλλες περιπτώσεις. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρει η πρωτοβουλία και συγχαίρω τον πρόεδρο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας και όλη τη Διδασκαλική Ομοσπονδία και τη διοίκηση που είναι παρόντες, διότι πρέπει επιτέλους το θέμα αυτό να λυθεί. Δεύτερον, πρέπει να υπάρξει ένα μήνυμα. Έχει νόημα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ρωτούν όλοι. Θα στηρίξει τα δικαιώματα των πολιτών. Ιδίω τώρα που πλησιάζουν και οι ευρωεκλογέ. Πρέπει να αποδείξει στην πράξη η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι υπάρχει, ότι λειτουργεί, και η βασική αρχή ποια είναι. Να εφαρμοστεί η νομοθεσία. Τι προτείνουμε λοιπόν. Πρώτον, να παραμείνει η αναφορά ανοιχτή. Δεύτερον, να στείλουμε επιστολή στο Υπουργείο Παιδείας και στο Υπουργείο Οικονομικών να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους και τρίτον, όπως είπε η Κομισιόν, να ενθαρρύνουμε την Κομισιόν να προχωρήσει σε έρευνα προκειμένου να ανοίξει φάκελος παραπομπής της Ελλάδος στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εάν δεν λύσει το θέμα. Δηλαδή, πρώτον, δεν προχωρήσει στη μονιμοποίηση των 22.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών δασκάλων και νηπιαγωγών και δεύτερον, να σταματήσει τώρα την παραβίαση των δικαιωμάτων τους, να έχουν τα ίδια εργασιακά δικαιώματα, τις ίδιες δυνατότητες προαγωγής με τους άλλους συναδέλφους τους. Ένας αναπληρωτής, εάν αρρωστήσει όπως σας το είπε ο πρόεδρος, μετά από 15 μέρες δεν έχει αναρωτική άδεια, τον απολύουν. Δεύτερον, παίρνει μισθούς και αυξάνονται αν θέλετε οι αμοιβέ του, λαμβάνοντα υπόψη την προϋπηρεσία, μέχρι τα 7 χρόνια. Ενώ οι υπόλοιποι μόνιμοι υπολογίζονται μέχρι και εργασία 40 ετών. Και αν σας φέρω και ένα παράδειγμα κύριε Πρόεδρε, δεν μπορούν να ασκήσουν και εκλογικά δικαιώματα. Εάν ένας αναπληρωτής δάσκαλο θέλει να είναι υποψήφιος σε ευρωεκλογέ, υποχρεώνεται από το ελληνικό δημόσιο να παρετηθεί από τη θέση του. Αν παρετηθεί όμω από τη θέση του, χάνει τα μόρια και επομένως την επόμενη χρονιά μπορεί να μην προσληφθεί. Αυτό που σας λέω το έθεσα υπόψη του Υπουργείου Εσωτερικών. Δηλαδή έχουμε πλήρη παραβίαση τη νομοθεσία. Επομένω, στηρίζουμε την αναφορά και επιμένουμε στο να παραμείνει ανοιχτή να στείλουμε επιστολή, όπως είπα, στο Υπουργείο Παιδείας και στο Υπουργείο Οικονομικών και να ζητήσουμε όμως από την Κομισιόν, αυτό είναι το βασικό, να επισπεύσει τις διαδικασίες ελέγχου και να παραπευθεί η Ελλάδα για διαχρονική παραβίαση. Διότι δεν αφορά μόνο αυτή την κυβέρνηση υπόθεση, αφορά τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Από το 1999 μέχρι σήμερα οι άνθρωποι αυτοί είναι σε ομοιρία. Υπάρχει εκπαιδευτικός ο οποίος δουλεύει 18 χρόνια και ακόμη είναι στον αέρα. Και να μην μας πούν ότι θα κάνει η κυβέρνηση προσλήψη στο μέλλον. Αυτό είναι μια καλή προοπτική. Εμείς θέλουμε εδώ και τώρα δικαίως των 22.000 συμπολιτών μας. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να δουν λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι ή όχι, και θέλουν να δουν την απόφαση τώρα, όχι μετά τις ευρωεκλογέ. Διότι διαφορετικά καταλαβαίνουν ότι δεν έχει νόημα να λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση αν δεν στηρίζει τα δικαιώματά τους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συγχαίρομαι και εγώ το Σωματείο των Εργαζομένων ε, Δασκάλων. Ε, ευχαριστώ και σε εσά, Πρόεδρε. Νομίζω ότι οι συμβάσει ορισμένου χρόνου στη δημόσια εκπαίδευση είναι μια μεγάλη πληγή, αλλά γενικά είναι μια ε, κοινωνική πληγή της φιλελεύθερης πολιτικής και αυτό στην Ελλάδα συμβαίνει από το 2001, όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι δουλεύουν σε αυτή την κατάσταση από το 2001. Αυτό σημαίνει ότι οι νέες γυναίκες και τα κορίτσια τα οποία θέλουν να κάνουν οικογένεια και να αγγίσουν παιδιά δεν έχουν δικαιώμα. Οι άνθρωποι που είναι άρρωστοι με καρκίνο δεν έχουν δικαιώμα για θεραπεία. Πώς? Γιατί μια θεραπεία καρκίνο είναι χρόνια και αυτοί δεν έχουν δικαίωμα πάνω από 15 μέρες αναρωτική άδεια. Φαντάζεστε σε τι κατάσταση εργάζονται αυτοί οι εργαζόμενοι και πόσο μεγάλη κοινωνική πληγή είναι μια παρόμοια φιλελεύθερη ρύθμιση. Έχουν δίκιο οι εργαζόμενοι και καταλαβαίνω ότι και εσείς μπορείτε να μπείτε στη θέση τους και να καταλάβετε τι βιώνουν. Όμως δίκιο έχουν σε αυτή τη φάση και αυτή η κυβέρνηση που έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια από ένα διάστημα κάπου προς το τέλος του μνημονίου και προσπαθεί να κάνει μια αρρύθμιση και να εντάξει με μια σκέψη δίκη όλους τους δασκάλους στην δημόσια εκπαίδευση. Αυτό σημαίνει ότι, όσο καταλαβαίνω, δεν είναι δυνατόν όλοι δεκάδες χιλιάδες να μπουν αμέσως στο σύστημα, αλλά θα υπάρχει ένας προγραμματισμός και μια προσπάθεια αυτό να συμβεί με τα χρόνια μπροστά. Προτείνω αυτή η αναφορά να μένει ανοιχτή, να υπάρχει ένας διάλογος και να ζητήσουμε στοιχεία από το Υπουργείο ακριβώς τι σκέφτεται να κάνει και να δούμε πώς θα είναι η εξέλιξη. Να κρατήσουμε την αναφορά έως να ολοκληρωθεί η εξέλιξη έως να καταχυρώσουν τα δικαιώματα των εργαζομένων στην εκπαίδευση. Thank much, Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίε και κύριοι, ε, η είναι στη διάθεσή μας για λίγα λεπτά ακόμα. Ε, ξεκίνησε κάπως δύσκολα η σημερινή μας συνεδρίαση. Ε, θα προσπαθήσω να συνοψίσω την κατάσταση. Η κατάσταση είναι απλή. Είναι σοβαρή η κατάσταση. Όλοι στηρίζουν την αναφορά αυτή. Θα παραμείνει λοιπόν ανοιχτή. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα δείξουν οι έρευνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και προς τον Υπουργό Εκπαίδευσης της Ελλάδας θα στείλουμε επιστολή και θα ζητήσουμε χρονοδιάγραμμα για την επίλυση του προβλήματος. Κύριε Μαριά. Πρόεδρε, συμφωνώ μαζί σας απλά. Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ μαζί σας απλά. Η επιστολή θα πρέπει να πάει στο Υπουργείο Παιδείας, όπως είπατε, αλλά και στο Υπουργείο Οικονομικών. Διότι το Υπουργείο Οικονομικών προσδιορίζει τα ποσά για τα οποία ε, πρέπει να καταβληθούν. Επίσης, θα πρέπει να το αποστείλουμε και στο Υπουργείο Εργασίας, διότι υπάρχει η άλλη πλευρά της αναφοράς, ότι μέχρι σήμερα παραβιάζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων για τις άδειες και όλα αυτά. Και στην Κομισιόν πρέπει να τη ζητήσουμε να επισπεύσει, να επισπεύσει την έρευνα to urge the Commission to investigate the Greek case διότι αν περιμένουμε μετά από χρόνια δεν θα έχει νόημα πρέπει άμεσα να ενεργήσει η Κομισιόν, να κάνει την ερευνά τη και να προετοιμάσει φάκελο παραπομπής κατά τη ελληνική κυβέρνηση. Διότι ένα θέμα είναι οι προσλήψει το οποίο, εγώ, το οποίο πρέπει, εμείς ζητούμε δικαίωση τώρα των 22.000. Προσλήψεις τώρα των 22.000 μονιμοποίηση, ένα, και να σταματήσει η παραβίαση των δικαιωμάτων τους. Τώρα, Ευχαριστούμε πολύ. Δεχόμαστε τις συστάσεις σας. Θα πάει επιστολή και στον Υπουργό Παιδείας και στον Υπουργό Οικονομικών. Σας ευχαριστώ πολύ. Λάβαμε την απόφαση αυτή και το Υπουργείο εργασία, γιατί μιλάμε και για εργασιακά δικαιώματα. Έχουμε τρία αρμόδια Υπουργεία. Το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εργασία. Λοιπόν, τρεις επιστολές θα αποσταλούν. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Διακόπτουμε αυτή τη στιγμή και θα συνεχίσουμε την όλη συζήτηση να λάβουμε και τις απαντήσεις στις επιστολές μας. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας και συνεχίζουμε τη συνεδρίασή μας στις 2.30. Ευχαριστώ.